και τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε την έκθεση Παμπλο Τζάλμπα Μπιντεγκάιν και Γκέρμπαν Γιάν Γκερμπράντι όσον αφορά την εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Τζάλμπα Μπιντεγκάιν. Έχετε το λόγο. Έχεις το λόγο, Παμπλο Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από ένα περίπου χρόνο, η Volkswagen ομολόγησε στον Οργανισμό Περιβαλλοντικής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι χρησιμοποίησε κάποια συστήματα αναστολής, defeat devices, για να περάσει τις δοκιμές καυσαερίων και να επιτύχει την έγκριση τύπου των αυτοκινήτων της στις Ηνωμένε Πολιτείε. Οπότε η πρώτη ερώτηση που θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι γιατί δεν αποκαλύφθηκε αυτό το σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να αποκαλύψει μια τέτοια εμβέλεια απάτη. Βέβαια δεν είναι εύκολο να βρούμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αλλά πολλοί παράγοντες ίσως θα μας βοηθήσουν να, το εξηγήσουμε. Εδώ είναι εμφανής μια έλλειψη της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια έλλειψη που οφείλεται σε ανεπαρκή ολοκλήρωση. Πιστεύω αναφίβολα ότι αν ήμασταν πραγματικά Ηνωμένα κράτη της Ευρώπης θα αποσοβούσαμε ένα τέτοιο σκάνδαλο, θα το αποτρέπαμε. Αν ήμασταν Ηνωμένα έθνη, Ηνωμένα κράτη της Ευρώπης, οι καταναλωτές μας, τα εκατομμύρια Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν καθημερινά τα γιοταχή τους, θα είχαν καλύτερης προστασίας. Επίσης πιστεύω ακράδαντα ότι αν είχαμε ένα ενιαίο δικαστικό σύστημα οι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμφίβολα θα έχουν καλύτερη προστασία. Υπάρχει όμως και άλλο στοιχείο που εξηγεί το πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Αναμφίβολα είχαμε μια ε, χαλαρή νομοθεσία επί Επιτρόπου Φερχόιγγεν ή μάλλον αφήσιμη σχετικά όριστη και έτσι εξηγείται πώς δεν καταφέραμε να αποκαλύψουμε αυτό το σκάνδαλο. Και έτσι έλαβε χώρα το σκάνδαλο, χάρη σε αυτή την σχετικά γενική νομοθεσία. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν την αυτοκριτική μας, γιατί ο Επίτροπος Φερχόγεν διαπραγματεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια νομοθετική πράξη που έδειξε τις, την ανεπάρκειά της και τις αδυναμίες της με το χρόνο. Στη συνέχεια ο Επίτροπος ε, Ταγιάννη προσπάθησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να προωθήσει μια φιλόδοξη νομοθεσία προκειμένου να μειωθούν τα οξύδια του αζότου, οι εκπομπές NOx. Και είχαμε αίσθηση των, συνέστηση των διαφορών. Και μάλιστα φάνηκε και από την έκθεσή μας ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ ε, των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και των δοκιμών στα εργαστήρια. Διαρωτόμαστε λοιπόν, κάναμε ότι έπρεπε τότε. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να κοιτάξουμε το μέλλον και αυτό περιμένουν οι καταναλωτές από εμά και από την εξεταστική μας επιτροπή. Να εξηχνιάσουμε την αλήθεια, αλλά να κάνουμε και προτάσεις για να υιοθετηθούν μέτρα ώστε να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων απατών. Πιστεύω αναφίβολα ότι όλοι οι συνάδελφοι θα συνεργαστούμε για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Και θα πρέπει όπω κάθε κρίση δημιουργεί ευκαιρίε και αυτή την κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας να την αξιοποιήσει η αυτοκινητοβιομηχανία για να προσαρμοστεί στην πολύ πιο απαιτητική πραγματικότητα του 21ου αιώνα για τα καυσαέρια. Πολύ πιο απαιτητική για την αναζήτηση νέων μορφών κινητικότητα. Επίση θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι τα έσοδα 12 εκατομμυρίων οικογενειών διακυβεύονται εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε αρκετά αυστηροί και να δείξουμε πυγμή όχι μόνο για να διασφαλίσουμε τα έσοδα αυτών των οικογενειών, αλλά κυρίως και πρώτα απ' όλα να τους εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Δεν έχει νόημα να αναγνωρίζουμε ότι γνωρίζαμε αυτή την απάτη. Θα πρέπει όμως να διαλευκάνουμε την αλήθεια και κυρίως να ατενίσουμε το μέλλον. Με ιδιαίτερη χαρά συνεργάστηκα με τον Ολαδό συνάδελφο και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία μας τους επόμενους μήνες και με τον κύριο Χερμπράντη και με τους υπόλοιπους και ηγητές και τους λοιπούς συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε εισηγητά. Ο λόγος στον άλλο εισηγητή. Στον κύριο Γκερμπράντη δίνουμε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον συνεισηγητή μου, τον κύριο Πάμπλο Ζάλμπα. Ήταν έξοχη δουλειά που έγινε μέχρι τώρα και προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί του τους επόμενους ε, μήνες. Αυτή η διάμεση έκθεση πρωταρχικά είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Υπήρχε λόγος γι' αυτό μόλις ξεκινήσαμε τις εργασίες μας, όμως υπάρχει και ένα πολιτικό σημείο σημαντικό. Καλούμε δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ταχύτερα και με καλύτερο τρόπο να συνεργαστεί με την Επιτροπή μας στην Εξεταστική αυτό έγινε όταν υθετήσαμε την ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτίωσε σημαντικά τη συνεργασία της και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η μέθοδος εργασίας. Μέχρι τώρα η Επιτροπή μας συνέλεξε, τι να τεχνικά στοιχεία θα έλεγα. Συζητήσαμε με εκπροσώπους αυτοκινητοβιομηχανίας, ε, παραγωγούς μηχανημάτων ελέγχου ρήπανσης, ε, ειδικού για το λογισμικό, πανεπιστημιακούς, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Κάναμε τεχνικής φύσεως εργασία μέχρι τώρα και ξεκινήσαμε τώρα το πολιτικό τμήμα της ε, έρευνας. Έγιναν ακροάσεις, ακούσαμε διάφορους επιτρόπους, ξεκινώντα από τον πρώην επίτροπο τον κύριο Δήμα, Πατοτσνίκ Φερχόγγεν και Ταγιάννη και χθε το βράδυ με τον παρόντα επίτροπο την κυρία Βιαρκόφσκα και Βέλα. Ε, θα είναι κρίσιμη και η συζήτησή μας όσον αφορά τα κράτη-μέλη και προσβλέπω στις ακροάσεις με εθνικούς υπουργούς τις επόμενες εβδομάδες και ειλικρινά καλώ τους υπουργούς εκείνους που δεν επιβεβαίωσαν θα παραστούν, τους παρακαλώ να το κάνουν. Η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία σημαίνει ότι και η εθνική υπουργοί είναι υπεύθυνοι για τη θέση που κατέχουν στην Ευρώπη Ακούσαμε την Αμερικανική EPA και τις Εθνικές Αρχές Εγκρίσεως Τύπου. Τι βρήκαμε μέχρι τώρα. Ανακαλύψαμε ότι είναι κάτι παραπάνω από μια υπόθεση που αφορά τη Volkswagen. Είδαμε ότι και άλλες αυτοκινητοβιομηχανές κλείνουν την τεχνολογία μειώσεως της ρήπανσης όταν η θερμοκρασία κατέβει κάτω από 17 βαθμούς ή μετά από 22 λεπτά που είναι πολύ κοντά στον κύκλο δοκιμών των 20 λεπτών, άρα το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο από τη Volkswagen και είναι κάτι που χρήζει περαιτέρω διερευνήσεως. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά επίσης όσον αφορά το ρόλο που έπαιξαν τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε ότι υπήρξε χαλαρή εφαρμογή και επιβολή της ευρωπαϊκής ε, νομοθεσίας και αυτό είναι κάτι που πραγματικά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συζητηθεί με τους εθνικούς υπουργούς. Ένα άλλο θέμα που διερευνούμε είναι γιατί χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να αναπτυχθεί αυτή η δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες οδήγηση. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έγγραφο εργασίας είπε ότι θα πετηθούν το πολύ δύο χρόνια για να αναπτυχθεί αυτή η δοκιμή και είδαμε ότι χρειάστηκαν πολλά περισσότερα χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί δεόντως. Τέλος, ένα χρόνο μετά το, την αποκάλυψη του σκανδάλου, ε, έχει περάσει από λοιπόν ένας χρόνος, έχουν γίνει πολλά έκτοτε, αλλά υπάρχουν ε, εκατομμύρια αυτοκίνητα με κινητήρα diesel που δεν συμμορφώνονται με τη σχήουσα νομοθεσία και είναι κάτι που το συζητήσαμε χθε με την Επίτροπο Μπιερκόφσκα και χαίρομαι διότι ακολουθεί μια στεναρή προσέγγιση. Περιμένουμε σε μερικές εβδομάδες διαδικασίες κατά παράβαση να ξεκινήσουν, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε προσεκτικά. Και η ανάκληση οχημάτων ε, βασίζεται πρωταρχικά επί εθελοντικής προσεγγίσεως. Προσβλέπω στους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του χρόνου, η, θα ολοκληρωθεί η έκθεσή μα και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα για ό,τι συνέβη κατά το παρελθόν, αλλά επίσης θα καταλήξουμε σε κάποια μαθήματα για το μέλλον και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι της ερευνάς μας. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά και τώρα το λόγο η Επίτροπος, η κυρία Μπιενκόφσκα έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και χαίρομαι που είμαι παρούσα Καταρχάς ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές για την εργασία τους. Είναι σχεδόν ένας χρόνος από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο Volkswagen και πάνω από έξι μήνες από τότε που η εξεταστική σας επιτροπή ξεκίνησε να εργάζεται και για όλους μας ήταν ε, μια περίοδος ε, έντονης εργασίας και για το Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας διαβεβαιώ ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να συνεργαστώ πλήρως και διαφανώς μαζί σας και δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω σε αυτή την οδό να συνεργάζομαι πλήρως με το Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες και μέχρι να λήξει η εργασία της Επιτροπής σας. Έκανα ό,τι μπορούσα για να απαντήσω σε όλες σας τις ερωτήσεις. Ξέρω ότι δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι, αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε και θα συνεχίσουμε. Είμαι πεπισμένη ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκαλυφθούν όλα τα στοιχεία και για να καταλήξουμε στα καλύτερα μέτρα ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως κράτη-μέλη ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος και ο κλάδος να είναι σύγχρονος και να αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις του για το περιβάλλον. Και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να είμαστε απόλυτα διαφανείς και να συνεργαζόμεθα. Και καλέσαμε τα κράτη-μέλη να διερευνήσουν αν υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί αλλίωση στα οχήματα που κυκλοφορούν στην επικράτειά του και να μα υποβάλουν έκθεση. Και τέσσερα κράτη-μέλη, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν υποβάλει τι εκθέσει. Αυτέ οι εκθέσει έχουν υποβληθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι και δημόσιε. Πρόσφατα, τέλη Ιουλίου, στείλαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια πρώτη επισκόπηση των εθνικών ερευνών, αλλά δυστυχώ δεν έχουμε την απόλυτη, την πλήρη εικόνα. Τα στοιχεία που μας έστειλαν τα κράτη-μέλη είναι ε, ανεπαρκή και θα χρειαστούμε και περαιτέρω τεχνική πληροφόρηση. Ε, προσωπικά και οι υπηρεσίες μου είμαστε απογοητευμένοι από την κατάσταση πραγμάτων. Χρειαζόμαστε αυτά τα τεχνικά στοιχεία για να μπορούμε να κάνουμε μία ανεξάρτητη αποτίμηση του τι συνέβη. Επέμεινα έναντι των κρατών μελών να μου αποστείλουν αυτά τα στοιχεία και θα επιμένω περαιτέρω στο μέλλον. Και παρακολουθώ και πώς προχωρούν οι εθνικές ε, έρευνες επ' αυτού. Κάτι τώρα για αυτούς τους μηχανισμούς αλλίωσης. Απαγορεύονται στην Ένωση. Εδώ και ε, πάνω από 18 χρόνια. 18 χρόνια! Και οι νομικές διατάξεις για αυτούς τους μηχανισμούς είναι σαφείς. Οι κατασκευαστές και όλες οι αρχές έγκρισης τύπου ποτέ δεν έθεσε να αμφιβόλο τους κανόνες αυτούς στην την εφαρμογή τους. Εάν δεν τους στηρούν, πρέπει να υπάρξουν επιπτώσεις. Γιατί παραβαίνουν τον νόμο. Και είμαι διατεθειμένη να επιβάλλω μια συνεπή εφαρμογή των κανόνων παντού στην ενία αγορά. Και οι υπηρεσίε μου και εγώ προσφερθήκαμε να δώσουμε πρακτικές οδηγίες στα κράτη-μέλη για το πώς να κάνουν τους ελέγχους εκπομπών κατά την έγκριση τύπου. Ελπίζουμε να υπάρξει λοιπόν συνεπής προσέγγιση σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Ξέρουμε ότι το κύριο πρόβλημα είναι η εφαρμογή του νόμου. Αυτό πρέπει να επιληθεί επιγόντως. Η παρούσα κατάσταση υπήρξε λόγω επικούς εφαρμογής και ανεπαρκούς επιτήρησης της αγοράς. Θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση. Θα υπάρξει ένα νέο σύστημα επιτήρησης με επικεφαλή στην Επιτροπή και αμοιβαίους ελέγχου μεταξύ κρατών μελών μαζί με ενωσιακέ κυρώσει. Όλα αυτά είναι ζωτικά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και για να επανέλθει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η οποία θίγει σοβαρότατα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της τον Ιανουάριο, τρέχοντος, και τώρα εναπόκειται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αποφασίσουν. Στο Συμβούλιο δεν έχουν καταλήξει σε θέση θα εργαστούμε ε, μέσω της ΙΜΚΟ, μέσω της έκθεσης του κύριου Ντόλτον για να προχωρήσουμε, αλλά και για να εγκριθεί η πρόταση όσο γρήγορα γίνεται. Η απροθυμία, θα έλεγα και αντίδραση στις αναγκαίες αλλαγές είναι αποθαρρυντική, για να μην πω απογοητευτική. Για να επιτύχουμε χρειαζόμαστε τη στήριξή σας, για να παραμείνει φιλόδοξη αυτή η πρόταση. Ελπίζω η εργασία της Επιτροπής ΕΜΙΣ να καταδείξει πόσο σημαντικές είναι οι προτινόμενες αλλαγές για το σύστημα έγκρισης τύπου των κρατών μας. Σας καλώ λοιπόν όλους να αντιμετωπίσετε το παρελθόν, αλλά όπως πάντα το βασικό είναι να ανοίξει ο δρόμος προς το μέλλον. Γιατί αλλιώς ε, παρά την τόσο έντονη εργασία μας δεν θα έχουμε απτά αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμεθα πλήρως μαζί σας τους επόμενους μήνες και για άλλη μια φορά η Επιτροπή χαιρετίζει την ενδιάμεση έκθεση και ελπίζω ότι θα επιτύχουμε και οι δύο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα θα ακούσουμε τις θέσεις των πολιτικών ομάδων. Πρέπει να ψηφίσουμε εγκαίρως. Ας μην χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη φάση τις γαλάζιες κάρτες αν θέλετε. Ο συνάδελφος Καρίν για το ΕΛΚ έχει το λόγο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Περάσαν έξι μήνε. Κάναμε πολλέ ακροάσει, ε, εμπειρογνωμόνων, ε, μαρτύρων, πανεπιστημιακών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, Μιλήσαμε με τον κλάδο, τους κατασκευαστές, τους αντιπροσώπους και με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή επιτρόπους, νυν και πρώην. Και τι μάθαμε, πώς είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση. Αυτό ήταν το ερώτημα. Πώς το κάναμε αυτό στην Ευρώπη. Για ιδεολογικούς λόγους είχαμε έναν βασικό στόχο που είχε να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Ήταν η μείωση του διοξιδίου του άνθρακος που εκπέμπεται. Και γι' αυτό επιχειρήσαμε να προωθήσουμε τους κινητήρες diesel και, την, και να επηρεάσουμε την συμπεριφορά των καταναλωτών. Αλλά αγνοήσαμε ένα παράγοντα. Οι κινητήρες diesel εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, αλλά πολύ περισσότερα οξύδια του αζότου πολύ περισσότερα. Το οποίο είναι ιδιαίτερη επιβλαβή για τη δημόσια υγεία. Το αγνοήσαμε αυτό. Αγνοήσαμε αυτή την παρενέργεια της πολιτικής μας. Αυτή την ιδιαίτερα επιβλαβή παρενέργεια. Έτσι λοιπόν οι κινητήρες για τα Euro 5 και 6 που ενεκρίθησαν το 2007 επεδίνωσαν το πρόβλημα. διότι οι εκπομπές σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης ήταν πολύ ψηλότερες από τις εκπομπές σε κέντρα τεχνικού ελέγχου και επιπλέον δεν υπήρχε ευρωπαϊκή ε, ρύθμιση αλλά ε, ρύθμιση σε επίπεδο κρατών μελών για τους ελέγχους και το βασικό λοιπόν για το μέλλον είναι να βλέπουμε όλα τα αποτελέσματα των πολιτικών μας και οι έλεγχοι να γίνονται σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης και να επηρεάσουν περισσότερο την συμπεριφορά των κρατών μελών. Σα ευχαριστώ για του Σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Η κυρία Βαντέμπτε έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπω είπε σωστά η Επίτροπο, πέρασε ένα χρόνο από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο τη Volkswagen και όλοι μείναμε να συγκλονιστήκαμε και από τη συμπεριφορά μια από τι μεγαλύτερε ε, ε, εμβληματικές ε, επικές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπάθησε να αυξήσει τα κέρδη της ε, εις βάρος των πελατών της που δεν γνώριζαν την κατάσταση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλά, πολλές αρχές εγκριστή που οι αγοράς, αρχές εποπτείας αγοράς που ανακάλυψαν αυτά τα θέματα, αλλά δεν επισημάνθηκαν δεόντω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για πρώτη εξεταστική επιτροπή τα τελευταία δέκα χρόνια και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κακοδιοίκηση, αλλά να δούμε και το φαινόμενο γενικά. Και η Επιτροπή εμείς θα πρέπει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά και στα ευρωπαϊκά προϊόντα βρισκόμαστε στα μέσα της πορείας μας, αλλά ανακαλύψαμε ότι όχι μόνο η Volkswagen και πολλές άλλες εταιρείες ε, αξιοποίησαν τα νομικά παραθυράκια, απενεργοποιώντας τα συστήματα ελέγχου των καυσερίων σε κανονικές συνθήκες οδήγησης. Και μετά από μία δεκαετία έχουμε πολύ περισσότερα καυσαέρια και εκπομπές ε, ε, επιζημιών αερίων και παραβιάσεις του νομικού μας πλαισίου. Και μάλιστα τα τζελοκίνητα έχουν τετραπλάσιες πενταπλάσιες εκπομπές από ό,τι παλιότερα και χαίρομαι για τη χθεσινή σας δήλωση κύριε Επίτροπε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι θα πρέπει να επαναπροσαρμόσουμε τα πράγματα και ε, αυτοκίνητα με συστήματα αναστολής καθημερινά εισέρχονται στις αγορές μας. Το να αφήνουμε να εκπέμπουν ε, θα αυξήσουν τη ρήπανση την ατμοσφαιρική τα επόμενα χρόνια. Επίσης, να επικεντρωθούμε στα κράτη-μέλη ε, και η εφαρμογή στο, σε εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ω πρόεδρος τη Επιτροπή Εμεί, τη Εξεταστική Επιτροπή, ελπίζω από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη, μέλη και εντό επιτροπή μα θα υπερκεράσουμε τι διαφορέ μα, τι πολιτικέ διαφορέ, και θα φανούμε σύσσωμοι στην προσπάθεια επίλυση αυτού του προβλήματο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για το ECR. Έχετε το λόγο συνάδελφε Χένκελ για 1,5 λεπτό. Κυρίε και κύριοι, πέρα από τι ε, εγκληματικέ ενέργειε και τα λάθη τη Volkswagen, η Επιτροπή έρευνα απέδειξε ότι απέτυχε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμη και ο Επίτροπος για τη Βιομηχανία, τότε ο Γκίντο Εφαχόγγεν, που είναι προκάτοχος της Επιτρόπου που είναι εδώ μπροστά μας, ε, παραδέχτηκε μετά από ερώτησή μου ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ήταν ιδιαίτερα σαφής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αμερικανικές προδιαγραφές για τις εκπομπές είναι πολύ πιο φιλόδοξες. Και όπως ήδη υπόθηκε, οι Αμερικανοί είναι εκείνοι απεκάλυψαν το σκάνδαλο, όχι εμείς οι Ευρωπαίοι. Άρα το συμπέρασμα, το μόνο λογικό συμπέρασμα πρέπει να είναι ότι πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαπραγματεύση για το TTIP να ζητήσει και την εναρμόνιση των ε, προδιαγραφών για τα ε, αυτοκίνητα και να υιοθετούνται ε, ανά περίπτωση τα υψηλότερα επίπεδα. Αυτό έχει τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Αυτό θα βοηθήσει την προστασία εκατομμυρίων πολιτών και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα εμποδίσει επιβλαβής για την υγεία τους εκπομπές και δεύτερον το κόστος ε, για την ε, εκπόνηση συστημάτων καυσαερίων θα μειωθούν και μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να καταδείξει πόσο μπορεί να είναι θετική. Με αυτόν τον τρόπο η Κομισιόν σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποδοχή του TTIP. Σας ευχαριστώ για την Άλντε. Συνάδελφε Καραντσόβα, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής ε, ε, εκτενή και αντικειμενική πληροφόρηση για το τι πραγματικά συνέβη. Οι ευρωβουλευτέ ε, θέτουν σαφεί ερωτήσει στην Επιτροπή για την αμέλεια που έδειξαν ή τι παραλήψει κρατομελών. Και θα έπρεπε να είχαμε ενημερωθεί δεόντω για την ύπαρξη και χρήση τέτοιων συστημάτων αναστολή. Κάτι που δεν συνέβη. Η εκπομπές ε, σε συνθήκες πραγματική οδήγηση θα έπρεπε να είχαν μετρηθεί και όχι μόνο στο εργαστήριο. Και αν ε, δεν αποκάλυπταν το σκάνδαλο οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, εμείς δεν θα το είχαμε εντοπίσει. Παρόλο που φάνηκε στην εμείς ότι το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια, γιατί τα αυτοκίνητα, αυτά τα διζελοκίνητα υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών, αλλά βρίσκουν τρόπους για να περάσουν παρόλα αυτά τους ελέγχους. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατείνεται ότι δεν υπήρχε ούτε παράληψη, ούτε κακοδιοίκηση. Κι όμως, δεδομένου των ατασταλιών που έγιναν, πολλά ερωτήματα έμειναν αναπάντητα. Χωρίς σαφείς απαντήσεις δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων καταναλωτών. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικό μα στόχο, η ανάκτηση αυτή τη εμπιστοσύνη. Εξού και η έκκληση μου προ του συζητητέ να εκπονήσουν μία έκθεση που θα είναι σαφή, ευανάγνωστη και φιλική προς τον αναγνώστη. Κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει από την έκθεση τι πραγματικά συνέβη και ποιος είναι ο υπέτειας ή ποιος είναι υπεύθυνος για την αποκάλυψη τέτοιων ατασταλιών και παρατυπιών. Θεωρώ ότι η έρευνα της Εξεταστικής Επιτροπής θα πρέπει να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα και να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από την έρευνα αυτή που να μετουσιωθούν στη νέα νομοθετική πράξη για την έγκριση τύπου και για τις μετρήσεις εκπομπών. Επίσης, η βιομηχανία που περιμένει την έκβαση των εργασιών της Επιτροπής ΕΜΗΣ έχει δημιουργήσει πάνω από 12 εκατομμύρια θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν χάσουμε και άλλο χρόνο, και αν κολυσιεργήσουμε περαιτέρω θα επιβραδύνουμε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Δυστυχώς δεν βλέπω κανέναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου εδώ. Μίζω σφάλμα. Γιατί όλα τα κοινωνικά θεσμικά όργανα θα πρέπει, κοινωνικά θεσμικά όργανα να βρουν απάντηση από κοινού. Ο κύριος Ηλικιώτης για 1,5 λεπτό για την ΚΟΥ. Έχετε το λόγο. Το Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πρώτη έκθεση που βάλει η Εξεταστική Επιτροπή περιορίζεται στην περιγραφή του προγράμματος εργασίας και δεν προβαίνει σε καμιά πολιτική εκτίμηση καθώ η έρευνα συνεχίζεται. Αυτό όμω δεν σημαίνει πω δεν έχουν ήδη εξαχθεί τα πρώτα συμπεράσματα. Αντιθέτω, μετά από πολλέ ακροάσει και μελέτη εσωτερικών εγγράφων, είναι πλέον ξεκάθαρο πω υπάρχουν σοβαρέ πολιτικέ ευθύνε. Τόσο οι εκτιμήσει του 2010, όσο και η μελέτη του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου τη Κομισιόν το 2013 επιβεβαίωσαν πω υπήρχε δυνατότητα αλλίωση των μετρήσεων κι όμω δεν λήφθηκε κανένα μέτρο. Η Κομισιόν γνώριζε για τη δυνατότητα απάτη, αλλά δεν έπραξε τίποτε με τη δικαιολογία ότι δεν γνώριζε συγκεκριμένε περιπτώσει. Και τα κράτη-μέλη, αν και είχαν ενημερωθεί, επίση δεν έκαναν κανέναν έλεγχο. Επίση, ενώ ήταν γνωστό πω οι μετρήσει εκπομπών είναι πολύ ψηλότερε σε πραγματικέ συνθήκε σε σχέση με τι τιμέ που καταγράφονται στα εργαστήρια, δεν ζητήθηκε να γίνονται έλεγχοι μόνο σε πραγματικέ συνθήκε δρόμου. Υπήρξαν λοιπόν σημαντικές παραλήψεις και από την κομισιόν αλλά και από τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και στην επιβολή κυρώσεων. ας πούμε όμως τα πράγματα με το όνομα τους τα κενά στην νομοθεσία οι ισχυρές πιέσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και το δίχτυ προστασίας των πολυεθνικών εταιριών οδήγησαν στο πολιτικό σκάνδαλο με τις μετρήσεις των εκπομπών. γιατί η απάτη της volkswagen δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Εμεί, αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε την έρευνα και θα ασκήσουμε περαιτέρω πιέσει. Θα συνεργαστούμε πάντοτε επικοδομητικά με του συζητητέ και του κοιοδησηγητέ για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Στόχο μα είναι να τερματιστούν όλε οι πρακτικέ που έχουν σαν στόχο το αθέμητο κέρδο σε βάρο τη δημόσια υγεία και του περιβάλλοντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Τούρμες για δυόμιση λεπτά εν ονόματι των Πρασίνων. Έχετε το λόγο κύριε Τούρμες. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο. Thank you. Ευχαριστώ. Πέρασε ένας χρόνος από το σκάνδαλο της Volkswagen. Είναι ένα σκάνδαλο όλη τη αυτοκινητομηχανίας. Απρίλιο-Μάιο του 2014 χέστον ΙΠΑ λαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία που δείχνουν διαφορές. Δεν γνώριζαν τίποτα για αυτές τις συσκευές αλλίωσης τι έκαναν οι Αμερικανικές αρχές τότε. Ζήτησαν από τη Volkswagen να απαντήσει το εξή. Μπορείτε να εξηγήσετε παρακαλώ τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της δοκιμής στο εργαστήριο και των υψηλών εκπομπών στην κανονική οδήγηση. Μη πρώτη συνάντηση, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη συνάντηση, πέμπτη συνάντηση. Η Volkswagen εψεύδεται συνεχώς. Μετά από 15 μήνες, το Σεπτέμβριο του 2015, αρχές των ΗΠΑ είπαν τελείωσε το παιχνίδι, η Volkswagen θα πρέπει να παραδεχτεί ότι διέπραξε ε, απάτη μεγάλης κλίμακας. Μετά η Volkswagen προσπάθησε να ανακαλέσει οχήματα στις ΙΠΑ. Ε, ε, να μία δράση, δεύτερη, τρίτη δράση ανακλήσεως. Οι αρχές των ΙΠΑ είχαν μία πλούστοτη ερώτηση. Μπορείτε να μας δείξετε ότι οι εκπομπές οξυδίων του αζότου με την, πληρούν την νομοθεσία μετά την ανάκληση δεν μπόρεσε να τα αποδείξει αυτή η Volkswagen. Καμία από αυτές τις δράσεις τους δεν ήταν αποτελεσματική. Μετά καταλήξε στην τρίτη πράξη. Αποζημίωση των καταναλωτών και τεράστια πρόστιμα για το μη σεβασμό της νομοθεσίας. Ο Ομπάμα και η κυβέρνησή του δεν έκανε τίποτα άλλο παρά τη δουλειά της. Έχεις μια βιομηχανία που εξαπατά και τελικά συλλαμβάνεται, πιάνεται στα πράσα. Τι κάναμε στην Ευρώπη είχαμε τις ίδιες πληροφορίες όπως και οι Αμερικανοί χρόνια πριν, το χειμώνα 2009-2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη δεν ρώτησαν ούτε μια φορά την Volkswagen, την εταιρεία. Δεν έθεσαν το ίδιο ερώτημα όπως οι Αμερικανοί. τι υπάρχει διαφορά μεταξύ των εκπομπών στο εργαστήριο και στην κανονική οδήγηση. Καμία δικασία για την παράβαση μέχρι σήμερα. Άρα συμμετέχει σε αυτή την ομερτά συνωμοσία σιωπή και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ίδια δράση ανάκληση τη Volkswagen που αρνήθηκαν οι Αμερικανικέ αρχέ τώρα έγινε δέκτη από την KBA. Δηλαδή ξανά εξαπατά τους καταναλωτές η Volkswagen με το επίσημο σήμα της γερμανικής κυβερνήσεως. Ερχόσαστε σήμερα χωρίς καμία δράση καμία προσπάθεια για ανάκληση. Γιατί δεν κινείστε επ' αυτού. Τρίτον θέμα είναι οι αποζημιώσεις. Καμία αποζημίωση. Λοιπόν, δηλαδή συνθηκολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον συνοψίζουμε, έρχεται η Επιτροπή Juncker. Δεν είναι αποκατασταθεί εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει δράση για την αποζημίωση, για την ανάκληση οχημάτων κλπ. Δεν μπορούμε λοιπόν με αυτή την στάση της Επιτροπής Γιούνκερ να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, κάτι που απαιτείται. Ευχαριστώ συνάδελφε Εύη για το EFTD, για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παρά τις ε, χαμηλές προσδοκίες για την Εξεταστική Επιτροπή, Γίνονται, συλλέγονται πολλά στοιχεία όμω μέσω των εργασιών τη Επιτροπή, που είναι χρήσιμα στοιχεία για να δούμε τις ε, και την αδιαφάνεια όσον αφορά την ιδιοδότηση των οχημάτων και τον έχω των εκπομπών του. Ένα σίγουρο πράγμα υπάρχει. Αυτές οι συσκευέ αλλίωση είναι απλώ η κορυφή του παγωβόνου του συστήματο. Δεν θέλω να επεκταθώ στην έκθεση, αλλά δράτω με τις ευκαιρία τη παρεμβάσεω στην Ολομέλεια για να πω δημοσία ότι έκθεση έρευνα όσον αφορά τα οχήματα Euro 5, τα δυσλοκινητήρα που πολλούνται στην Ιταλία, έκθεση που έκανε το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών της Ιταλίας, είναι μια προσβολή στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αυτού του Κοινοβουλίου και κυρίως σοβαρά προσβλητικό έναντι των Ευρωπαίων πολιτών που αξίζουν διαφάνεια, σοβαρότητα από πλευράς των θεσμικών οργάνων. Η έκθεση είναι ατελής ε, οι έρευνες για τα 15 οχήματα που αναφέρονται στην έκθεση ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες ε, όσον αφορά τις διάφορες ομάδες οχημάτων. Τα αυτοκίνητα Fiat εξετάζονται στα εργαστήρια Fiat της Τωρίνα και άλλα οχήματα στα αρχεία της CNR. Χάνονται τα ίχνη κάποιων μοντέλων Jeep και Fiat, εξαφανίζονται από τις γραφικές παραστάσεις και από τους πίνακες. Υπάρχουν μόνο μοντέλα για τα ΕΠΑ, υπάρχουν οι μεγαλύτερε υπόνοιε όπου διαθέτουν αυτέ ε, του μηχανισμού αλλίωση και μηχανισμούς που κλείνουν μετά από 22 λεπτά, 2 λεπτά μετά τον κύκλο δοκιμής της έγκρισης τύπου και έχουμε και ένα άλλο μοντέλο που στις δοκιμές εμψυχρό ε, είχε ε, εκπομπή οξυδίου του τρεις φορές παραπάνω από το κανονικό. Γίνεται αδέξιος τρόπος ε, να καλύπτουν οι πραγματικές τιμές των εκπομπών των Fiat. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε ότι αυτή η έκθεση είναι προσβολή και προς την έκθεση Εξεταστικής Επιτροπής και προς το Κοινοβούλιο και προς πολίτες. Ευχαριστώ συνάδελφε Πρέτσελ για το ΕΝΕΦ. E Έχετε το λόγο για δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πέρα από το γεγονός ότι η Volkswagen προφανώς ε, παρεύει τον νόμο, μάθαμε και διάφορα άλλα μέσω των ακροάσεων των τελευταίων μήνων διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι φαίνεται, δεν ασκούσε επαρκώς τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου και δεν είχε επαρκείς δυνατότητες ελέγχου και τις δυνατότητες, τις λίγες δυνατότητες που είχε, από ό,τι φαίνεται δεν τις καταλάβαινε και δεν τις εφήρμοσε σωστά. Κυρία Μπιενκόφσκα, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχουν ε, ε, πολλές ενδείξεις, όχι μόνο φήμες, ότι υπήρχαν τέτοια προβλήματα όχι μόνο με την Volkswagen, αλλά και από άλλες εταιρείες. Και ξέρετε ότι έχετε όλα τα τεχνικά στοιχεία. Θα μπορούσατε να έχετε ζητήσει όλα τα τεχνικά στοιχεία, όχι μόνο από τη Volkswagen, από άλλε εταιρείε. Και δεν το κάνετε. Και ακόμη δεν μα εξηγήσατε τι θα κάνετε έναντι των κρατών που είναι υποχρεωμένα να σα στείλουν τα τεχνικά στοιχεία και δεν το κάνουν. Δεν έχετε συστήματα ελέγχου τη ποιότητα για την εφαρμογή του νόμου. Και επιπλέον, συνάδελφοι, αν θέλουμε η νομοθεσία μας να λαμβάνεται σοβαρά, αν θέλουμε να υπάρχουν ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, τότε πρέπει να υπάρχουν τα συστήματα ελέγχου της ποιότητας. Αντί για όλα αυτά, βασιζόμεθα στις πληροφορίες από αμερικανικές υπηρεσίες. Και ίσως, ίσως, να παίζει ρόλο σε αυτό και η διαφορετικότητα των οικονομικών συμφερόντων Ένωσης ΗΠΑ. Δεν πρέπει λοιπόν να υπολοιπόμεθα των Αμερικανών και να ακολουθούμε αυτά που μας λένε. Πρέπει να έχουμε ανεξάρτητη πηγή πληροφόρησης και αποτίμησης. Δεν είναι δυνατόν η Volkswagen να πληρώνει 15 δις αποζημιώσεις στις ΗΠΑ και εδώ τίποτα. Πρέπει να γίνουν και περαιτέρω κατασκευαστές. Αυτή η τελευταία παρέμβαση των πολιτικών ομάδων, συνάδελφε Γκίζε, και έχετε το λόγο για δύο λεπτά και καλώ του συναδέλφου να σέβονται το χρόνο που διατίθεται, διότι έχουμε ένα πρόβλημα με τι ψηφοφορίε που ακολουθούν. Πρέπει να ξεκινήσουμε έγκαιρα τι ψηφοφορίε, σύμφωνα με το ωράριο. Συνάδελφε Γκίζε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Συνάδελφοι. Έχουμε φτάσει στο εμίχρονο στις σημαντικές εργασίες της Επιτροπής για τα καυσαέρια και έχει γίνει σημαντική τεχνική εργασία. Είμαι πεπισμένο ότι ήδη έχουμε επιτύχει κάποιες πρόοδους θα πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία υψηλή ποιότητα, την τεχνική εργασία και πρέπει να δούμε και τι πολιτικέ επιπτώσει. Ορισμένοι συνάδελφοι λένε ότι η Κομισιόν και κάποιοι επίτροποι θα έπρεπε να ξέρουν για αυτού του μηχανισμού. Αλλά καμία απόδειξη δεν έχει δοθεί ούτε τις τελευταίες εβδομάδε. Παρά το ότι υπόθηκε ότι η Επίτροπος Ποτότσνικ έπρεπε ή μάλλον είχε στείλει μια επιστολή στον συνάδελφο του Ταγιάννη, αλλά δεν έχουμε δει καμία τέτοια επιστολή, άρα όλα αυτά είναι αναπόδεικνα. Θα ήταν ε, ε περίεργο για το ίδιο ο Ποτότσνικ είπε ότι δεν είχε υπόψη για τέτοιου μηχανισμού. Πώ είναι να τον έχει αποστείλει τέτοια επιστολή. Να δούμε τώρα πώ θα πάει το δεύτερο εμίχρονο. Εγώ προτείνω για αυτό το δεύτερο εμίχρονο να σταματήσουμε αυτά τα πολιτικά παιχνιδάκια. Και αντί γι' αυτό να βελτιώσουμε την νομοθετική διαδικασία στην Κομισιόν η διαφορά μεταξύ των μετρήσεων ε, σε συνθήκες εργαστηρίου και κυκλοφορίας ήταν γνωστές οι διαφορές αυτές για τις εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου. Πρέπει λοιπόν και το Κοινοβούλιο να συμπεριληφθεί στου νέου κανονισμού, στο καθορισμό των νέων κανονισμών. Και δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε τόσο πολύ για να καταλήξουμε σε αυτού του νέου κανονισμού για τι εκπομπέ. Συμφωνούν όλε οι πολιτικέ ομάδε επ' αυτών. Ελπίζω να επιτύχει η Επιτροπή μα πρώτα απ' όλα να παραμείνει επί τη ουσία, να αποφύγει τη μικροπολιτική και επιπλέον να είναι σαφέστερη η διατύπωση τη νομοθεσία στο μέλλον που να μην επιτρέπει απάτε. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Ντάντς, έχει το λόγο για μισή λεπτό. Ε, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως αναφέρθηκε, πρέπει να αποτιμήσουμε το έργο της Επιτροπής ε, της Εξεταστικής. Τι απεκάλυψε. Ακούσαμε ήδη ότι ελήφθη μια απόφαση κατά το παρελθόν να κινηθούμε προς ένα τομέα που οδηγήθηκε σε υψηλότερες εκπομπές οξυδίων του Θέλαμε να μειώσουμε τι εκπομπέ του εξωτερικού άνθρακο, αλλά είχε αυτή την παράπλευρη απώλεια. Υπήρχε έλλειψη γνώση και στοιχείων όσον αφορά τα αποτελέσματα που έχει ο διζελοκινητήρα στη δημόσια υγεία. Ένα κομμά, τμήμα για τον οποίο, μια ένα αίτιο για τον οποίο δεν είχαμε τα στοιχεία ήταν ότι υπήρχαν πάρα πολλές λεπτομέρειες που έπρεπε να αποκαλυφθούν και κανένας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες. Κατηγούνται κάτι μέλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί τα κράτη-μέλη, η αυτοκινητοβιομηχανία ε, περνά από διάφορα κενά της νομοθεσίας και ωφελείται από την νομοθεσία και ξεφεύγει από το δίκτυο. Τι ανακαλύψαμε μέχρι τώρα λοιπόν, ότι υπάρχει φοβερή διαφορά όσον αφορά την ερμηνεία τη κείμενη νομοθεσία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο σε αυτό που λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα πορίσματα τη Εξεταστική Επιτροπή, ώστε η επόμενη νομοθεσία να μην ε, έχει τα ίδια σφάλματα και τα ίδια κενά και δυνατότητες για ε, αμφίσιμη ερμηνεία. Πρέπει να είναι σαφή η νομοθεσία. Τέλο, θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφου από όλο το πολιτικό φάσμα. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να μην γίνει ένα πολιτικό παιχνίδι δεξιά και αριστερά, διότι το χωστούμε στου κατανοτέ τη Ευρώπη και την τομέα τη δημόσια στην Ευρώπη. Να πετύχουν σωστά αποτελέσματα. Συνάδελφε Ντεμεσμάκερ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ Είμαι υπέρ της ενδιάμεσης έκθεσης της Εξεταστικής Επιτροπής εμείς ε, και ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής και παρόλο που είναι πρόημο να αντιλήσουμε κάποια οριστικά συμπεράσματα, μπορούμε κάποια ενδιάμεσα συμπεράσματα να ε, αντιλήσουμε. Για παράδειγμα ότι οι δοκιμές γίνονται σε εργαστήριο και όχι σε πραγματικές ηθίκες οδήγησης. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε πιο αποτελεσματικές δράσεις για να γίνει σεβαστή η νομοθεσία, να τηρηθούν οι κανόνες, να προστατεύσουμε την ανθρώπινη υγεία και επίσης να γεφυρώσουμε αυτό το, τεχνικό χάσμα γιατί υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογίες για να γίνουν σεβαστά τα όρια των καυσαερίων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και όχι μόνο τον, του διοξιδίου του άνθρακα αλλά και ε, των οξυδιών αζότου. Η νομοθεσία απαγορεύεται στήματα αναστολή, αλλά δυστυχώ υπήρχαν παραθυράκια που επιτρέπουν την περιστασιακή απενεργοποίηση τέτοιων μηχανισμών και επίση εξαρτάται και από την θερμοκρασία. Απενεργοποιούνται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Ο τελικός χαμένος είναι και ο καταναλωτής. Οι βασικές μας προτεραιότητες είναι να αποκαλύψουμε την πραγματικότητα, να προτείνουμε λύσεις για το μέλλον και να αξιοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές όπως στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Τόρβαλτς, παρακαλώ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την Επίτροπο Μπιανκόφσκα. Καλύτερα να μιλήσω ειδικά για να με καταλάβουν και οι συμπολίτε μου στη Σουηδία. Πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση, αλλά μας έφερε και σε δύσκολη θέση και σε αμηχανία, γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν σαφείς κανόνες και οι καταναλωτές, οι πολίτες ε, ε, δικαιούνται αποζημίωση από τη Volkswagen ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια και έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία αυτή τα απαγορευμένα συστήματα αναστολής ή αλλίωση των αποτελεσμάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάσταση είναι διαφορετική. Όχι μόνο έχουμε τέτοια συστήματα αλλίωση αποτελεσμάτων στα αυτοκίνητα μας, αλλά δυστυχώς και οι επιδόσεις μας ε, είναι πενιχρές και έγινε και μεγάλη χειραγώγηση με αποτέλεσμα να μένουν απληροφόρητοι οι καταναλωτές. Κάτι που δείχνει ότι δεν είναι υπέτεια μόνο η Volkswagen για το σκάνδαλο αυτό. Υπάρχουν και άλλες ε, υπεύθυνε αυτοκινητοβιομηχανίες. Θα πρέπει να ενημερώνεται ο καταναλωτής. Είναι σημαντικό για να έχει εμπιστοσύνη στα προϊόντα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό που αποδείξαμε, ότι δεν ήταν σωστή μέχρι τώρα η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν συνεχιστεί μια τέτοια κατάσταση, θα φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν θα αποζημιωθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες για τις ε, ζημίες που υπέστησαν για ένα ελαττωματικό προϊόν που αγόρασαν και που συμβάλλει στη ρήπαση του περιβάλλοντος. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να βοηθήσουμε τους καταναλωτές. Συνάδελφε Κίλωνεν, για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι η μείωση των εκπομπών. Στην κυκλοφορία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ φιλόδοξη. Ονειρευόμαστε ε, κυκλοφορία με σχεδόν μηδενικές ε, εκπομπές όμως ε, τελικά πρέπει να αποφύγουμε τη μεγάλη κερδοφορία των εταιριών. 400.000 ε, θάνατοι προξενούνται το χρόνο από τις εκπομπές των ε, αυτοκινήτων. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα του περιβάλλοντος, να ανταποκριθούμε στο στόχο. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Από την πλευρά της αυτοκινητοβιομηχανίας λοιπόν θα πρέπει να αποδεχτεί η αυτοκινητοβιομηχανία τις ευθύνες της. Από την πλευρά μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εργαστούμε ούτω ώστε οι εκπομπές να ελέγχονται σωστά και τα μέτρα να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Θα πρέπει λοιπόν να αντλήσουμε τα μαθήματά μας από το παρελθόν και το σκάνδαλο. Για ένα λεπτό και έχετε και εσείς το λόγο κύριε Κάουτ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα. Νομίζω ότι βλέποντας αυτά που μαθήσαμε από την Επιτροπή Εξεταστική, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λένε οι τεχνικοί εμπειρογνωμόνες, ότι δεν υπάρχει τεχνικός λόγος για να σβήσει η αδίποτε τεχνολογία μειώς εκπομπών. Δεν χρειάζεται για την προστασία των κινητήρων κάτι τέτοιο. Γνωρίζουμε όμως ότι Όλες σχεδόν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, όλες χρησιμοποιούν λογισμικό για να σταματήσει η λειτουργία της τεχνολογίας. Μόνο η Volkswagen ε, καταδικάστηκε για τη χρήση των συσκευών αυτής αλλίωση. Η Fiat κλείνει τον μηχανισμό μετά από 22 λεπτά ή άλλη παραγωγή αυτοκινήτων κάτω από 17 βαθμούς. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Καμία άλλη μάρκα αυτοκινήτων δεν κατηγορείται για τη χρήση μηχανισμών αλλίωση. Χρειάζεται κατεπίγοντος δράση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. όπω μιλάμε, ε, ακόμα κυκλοφορούν αυτοκίνητα που ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα. Πότε θα γίνει συντονισμένη ανάκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο ώστε τα βρώμικα οχήματα να φύγουν από την κυκλοφορία κατά του τους δρόμους μας. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Έλμερ, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω καταρχάς Συγχαίρω τους συναδέλφους διότι η συζήτηση όπως την ακούω είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από ότι η ενδιάμεση έκθεση που υποστηρίχθηκε ε, α, ομόφωνα από την Επιτροπή παράξενη έκθεση. Της λείπει το περιεχόμενο θα έλεγα, σχεδόν εντελώς. Ε, είναι ομφαλοσκόπηση στο έγγραφο. Στην παράγραφο 1 ζητά η Επιτροπή τον εαυτό της να εκπληρώσει την εντολή της. Αυτό φαίνεται παράξενο, μια ταυτολογία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περισσότερη συνεργασία. Όμως έχω πρόβλημα με μία λέξη της εκθέσεως. Είναι μία ύβριση παράγραφος 4 με ανέβεια. ζητά από τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να αναλάβουν κάποιες δράσεις. Δεν έχει καμιά δουλειά αυτό το κοινοβούλιο, ούτε η προσωρινή επιτροπή αυτού, να απαιτήσει από κυρίαρχε κυβερνήσει να αναλάβουν οποιαδήποτε δράση. Αν επικρατούσε η ευγένεια, αν ζητούσε αντί να πετύχει η Επιτροπή, τότε θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την έκθεση. Όσοι έχει, φοβούμαι ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Ζακ, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαιρετίζω τι εργασίε τη Επιτροπή μα που προσπαθεί να αποκαλύψει σε κάθε λεπτομέρεια τι ελλείψει ε, του κλάδου και τη Επιτροπής όσον αφορά του ελέγχου των καυσαερίων. Όμως οι εργασίες μας ασχολούνται με τεχνικά θέματα και παραμελούν το θέμα ότι τα προβλήματα της Volkswagen είναι στα πλαίσια ενός οικονομικού πολέμου ε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος θέλει να ε, σκοτώσει το σκύλο το κατηγορεί ότι έχει λύσα. Ε, έχουμε προβλήματα εδώ και ορισμένα χρόνια με τα οξύδια του αζότου ε, λόγω των κινητήρων δίζελ ενώ οι Αμερικανοί που προτιμούν τους κινητήρες βενζίνης ε, έχουν άλλη πολιτική. Πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί, πιο πολιτικοί. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Μπέλετ. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ήβο. Uh, uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Είμαστε στα μισά της ε, εργασίας της Επιτροπής αυτής και νομίζω ότι όπως υπόθηκε έχουμε μια καλή εικόνα ε, του τι ε, πήγε στραβά και πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι μηχανισμοί αλλίωσης και τι πρέπει να κάνουμε για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Υπάρχει κοινή ευθύνη, κυρία Επίτροπη. Νομίζω ότι το είπαμε σαφώς χθες στην ακρόαση μαζί σας. Κατεδείχθη σαφώς. Κανείς Ούτε εμείς ως Κοινοβούλιο δεν είχαμε πλήρη εικόνα της κατάστασης. Έπρεπε λοιπόν να επαρρυπνήσουμε πολύ περισσότερο για να ε, εξακριβώσουμε τη χρήση αυτών των μηχανισμών. Και ορισμένοι ομιλητές τόνισαν ότι και οι εθνικές αρχές δεν έλεγξαν επαρκώς, γιατί αυτές οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας την οποία εγκρίναμε από κοινού όλα τα 28 κράτη-μέλη και εμείς ως Κοινοβούλιο. Άρα, κύριε Επίτροπε, ε, βασιζόμεθα σε εσά. Εσείς έπρεπε να ελέγχετε τη διαδικασία ελέγχων και τη σωστή εφαρμογή, όπως είπε ο κύριος Χέλμερ. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζει ομοιόμορφα τους κανόνες. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική αυτή η έλεγχη. Διότι η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει όχι μόνο τα καλύτερα, αλλά και τα πιο βιώσιμα αυτοκίνητα, βιώσιμα για το περιβάλλον δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε στην πρωτοπορία αυτών των καθαρών τεχνολογιών. Τα 18 ε, μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο πρέπει να τηρούνται. Πρέπει λοιπόν να, να πιέσουμε τον κλάδο για να καταστεί σαφές ότι πρέπει να βάλουν πιο ψηλή ταχύτητα στις προσπάθειές τους. Γιατί μας απογοήτευσε όλους και απέτυχε και δεν σεβάστηκε και τις ανάγκες των καταναλωτών. Πρέπει λοιπόν το κοινοβούλιο μας να πιέσει όπως πρέπει ούτω ώστε να επανέλθει αυτή η εμπιστοσύνη προς τους καταναλωτές. Αυτό πρέπει να το κάνουμε μόνο με φιλοδοξία και διαφάνεια. Κοιτάξτε συνάδελφε, υπάρχει γαλάζια κάρτα για σας. Ε, δέχεστε. Συνάδελφε Φρουτσούλη, θέστε το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, καλωσορίζω την ομιλία σας και, θα ήθελα να υπογραμμίσω, υπογραμμίσω ε, την ανάγκη σωστής μεθοδολογίας και διαφάνειας της μεθοδολογίας ε, ε, της, Επιτροπής, της Εξεταστικής Επιτροπής εμείς. Πώς πιστεύετε ότι η Επιτροπή εμείς μπορεί να συμβάλλει, όπως είπατε, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και να εξασφαλίσει ε, την αποτροπή τέτοιου είδους σκαδάλων στο μέλλον. Ευχαριστώ για την ερώτηση, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δημοσίευση όλων αυτών των πληροφοριών. Θα πρέπει να είναι προσιτές στο κοινό όλες οι πληροφορίες. Όπως είπε η ε, κυρία Επίτροπος, κάποια έγγραφα που αρχικά είχαν κριθεί εμπιστευτικά τελικά θα γίνουν προσιτά στο κοινό. Επίσης, ε, να υποβάλουμε προτάσεις για την έγκριση τύπου και τι ε, κανονικέ ήθικες οδήγηση. Ελπίζω οι σχετικέ νομοθετικέ διατάξει να θεσπιστούν το συντομότερο δυνατό μετά από συμφωνία με το Συμβούλιο για να γίνουν νομοθεσία. Η κυρία Ρεβό Νταλόν Ντονφό. 1,5 λεπτό, Χριστίνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, είναι δύσκολο να εκπονήσει κανεί νομοθεσία για να φροντίσει, να καθορίσει πώ πρέπει να γίνεται η οδήγηση των οχημάτων, προστατεύοντα συγχρόνω την υγεία όλων μα. Πρέπει να σεβόμαστε του κανόνε βάσει της οδήγησης στους δρόμους και όχι βάσει της οδήγησης σε εργαστήρια όπου δεν υπάρχουν ούτε καθίσματα, ούτε θέρμανση, ούτε κλιματισμός. Δέκα χρόνια χρειάστηκαν για να φτάσουμε εκεί και παρόλα αυτά φτάνουμε με έναν δείκτη συμμόρφωσης 2,5. Αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο να φροντίσουμε να τηρούνται οι κανόνες, να τους ελέγχουμε και να επιβάλλουμε κυρώσεις. Σήμερα η κατάσταση είναι τέτοια που οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν πια, γιατί από αυτούς απαιτούμε να τηρούν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δυστυχώ όμω η αλυσίδα ελέγχου και κυρώσεων δεν λειτουργεί ούτε καν όταν πρόκειται για τη δημόσια υγεία. Η εικόνα λοιπόν τη Ευρώπη και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι κάκιστη και δεν είναι προ όφελο κανενών μα. Επειδή ακριβώ είμαι πεπισμένη Ευρωπαία και επειδή πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει το πολιτικό οικοδόμημα μέσα στο οποίο βρίσκεται, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Τα σκάνδαλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί αν όλε οι διαφερόμενε πλευρέ είχαν τηρήσει τον νόμο. Τίποτα άλλο, να είχαν τηρήσει τον νόμο αποτελεσματικά όμω. Έφτασε πια η στιγμή να υπενθυμίσουμε τι θέσει μα και να εξηγήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή για να υποστηρίξει το γενικό συμφέρον. Αυτό που διακυδεύεται εδώ δεν είναι να τα βάλουμε με τη βιομηχανία, ούτε βέβαια και να καλύψουμε αυτού οι οποίοι έθεσαν την οικονομία πάνω από άλλε αρχέ. Όχι. Αυτό που διακυδεύεται εδώ είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των πολιτών. Είναι να έχουμε μεταφορές πιο καθαρές, να σεβόμαστε τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, Προστατεύοντα όμω τι θέσει απασχόληση, με δύο λόγια, πρέπει να φροντίσουμε για μια βιώσιμη ανάπτυξη προ όφελο όλων. Και αυτό είναι και το κίνητρό μου ω μέλο τη Επιτροπή ΕΜΗ από την πλευρά των Σοσιαλιστών και αυτό είναι και το κίνητρό μου που βρίσκομαι εδώ σε αυτή τη θέση ω Ευρωβουλευτή. Ευχαριστούμε, κύριε Ντάλτον. Ευχαριστώ. λεπτό. Εδώ και ένα χρόνο ανακαλύψαμε ότι η Volkswagen παραπλάνησε του κατόχου αυτοκινήτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και έκτοτε τι έχει γίνει, Πώ έγινε αυτό χωρί να το έχουν δει οι ρυθμιστέ, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Κανένα σύστημα δεν είναι 100% σίγουρο, αλλά το βασικό είναι να το κάνουμε όσο δυνατόν πιο δύσκολο να παραπλανήσει κανεί του αγοραστέ και να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν. Τώρα έχουμε κάποιου κανόνε δοκιμών έτοιμου, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και έχουμε και κάποιε προτάσει τη επιτροπή, που είναι επίση σημαντικό. Πρέπει το συντομότερο δυνατόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Να έχουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα από την Εξεταστική Επιτροπή και να να έχουμε την τελική της έκθεση του χρόνου. Επίσης, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν την νομοθεσία, όπως μας είπε και χθε το βράδυ η Επιτροπή η Volkswagen να παραπλάνησε όλα τα κράτη, όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Χρειαζόμαστε σωστά σύστημα, σωστή εφαρμογή στα κράτη-μέλη και σωστή εποπτεία σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί και αν δεν μπορούμε να το παρέχουμε αυτό στου καταναλωτέ, θα είναι ει βάρο των καταναλωτών και του περιβάλλοντο. Ευχαριστώ. Κύριε Φαρία, δύο λεπτά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλα προβλήματα ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα στις πόλεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία στους δρόμους. Ε, πολύ μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων πολιτών εκτίθεται στις συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρήπανσης που αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Ε, πάνω από 70.000 άνθρωποι πεθαίνουν ε, κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των υψηλών επιπέδων ε, οξυδίων του αζότου στην ε, ατμόσφαιρα. Βασική πηγή είναι τα, η εξατμίσεις των αυτοκινήτων για αυτά τα αέρια στις αστικές περιοχές. Εμείς λοιπόν με την ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει κάπως να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν λειτουργήσε καλά αυτό το σύστημα. Φαίνεται να υπάρχει ε, μια ιδιαίτερη έμνοια προς την ε, οποιαδήποτε είδος βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας ε, δήθεν υπέρ των αυτοκινητοβιομήχανων. Ε, είναι, ότι πρέπει να αγωνιστούμε υπέρ τη βιομηχανική πολιτική. όμως όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην τεχνολογική καινοτομία και να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των πολιτών για καλύτερη ποιότητα ζωής της πόλη. Ε, θα πρέπει να στηρίξουμε τις πιο βιώσιμες ε, δημόσιες μεταφορές και την ηλεκτρική κινητικότητα που είναι πιο καθαρή και πιο φθηνή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, αυτά, στις, αυτά τα μέσα. Είναι ντροπή να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα όσον αφορά αυτή την απάτη για τις, τους ρήπους. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα όπως και οι Αμερικανοί ε, για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών. Θα είναι σημαντικό που δημιουργήθηκε αυτή η Επιτροπή Έρευνα. Είναι το, το μήνυμο λοιπόν που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να είναι πολύ επιμελή στη συνεργασία τη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αναζήτηση τη αλήθεια. Θα πρέπει να δούμε τι θα αλλάξει ώστε να υπάρξει διαφορετικό τρόπο ελέγχου τη εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πρώτη να είναι οι πολίτε. Δεν ίσχυσε όμω αυτό στη διάρκεια αυτή τη διαδικασία και δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε. Ε, κυρία για λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, αν κανείς δεν θέλει να μάθει την αλήθεια, τι κάνει, φτιάχνει μια εξεταστική επιτροπή. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια αποφάσισε να δημιουργήσει αυτό το μέσο, την εξεταστική δηλαδή επιτροπή, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να συνεργαστεί. Βρίσκει ένα σωρό άλοθη από την αυτοκινητοβιομηχανία κλπ. Η Εξεταστική Επιτροπή θέλει να βρει τι, αυτά τα οποία ήδη γνωρίζουμε. Το σκάνδαλο ήταν γνωστό το τι γινότανε δηλαδή, όλοι το ξέρανε, απλώς το κρύβανε, δεν το λέγανε. Και τώρα είμαστε αντιμέτωποι με την αντίσταση αυτών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και αυτών οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν με αλαζονικό τρόπο και μας έκρυψαν την αλήθεια. Θέλω να ευχαριστήσω παρόλα αυτά την Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής και όλους τους συναδέρφους. Φαίνεται ότι μπορούμε να βρούμε τελικά τις αιτίες του σκανδάλου αυτού. Ευχαριστούμε κυρία Ντελή. Ένα λεπτό. Καρίν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επέτροπη. Το σκάνδαλο Volkswagen ξέσπασε πριν από ένα χρόνο. Το σκάνδαλο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και τώρα ένα χρόνο μετά από αυτήν την φοβερή απάτη όσον αφορά τις δοκιμές για τις εκπομπές Τίποτα άλλο δεν έχει γίνει εκτό από την Εξεταστική Επιτροπή. Κανένα μέτρο δεν υιοθετήθηκε ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από τι χώρε μέλη για να τηρούνται τι οι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ για την προστασία του πολίτη και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Εδώ και ένα χρόνο δηλαδή αφήνουμε τον Ευρωπαίο πολίτη να τον ξεγελάνε, ενώ οι Αμερικανοί παίρνουν πίσω τα λεφτά τους. Εμείς τελικά τι κάνουμε, ρηπαίνουμε τους δρόμους μας και δεν κάνουμε τίποτα άλλο είπατε ναι ε, διαδικασίες ε, παραβάση κατά κάποιων χωρών. Είναι ένα πρώτο βήμα. Αλλά κατά τα άλλα τι περιμένετε. Η γαλλική κυβέρνηση προστατεύει τη Ρενό η οποία είναι από αυτούς που ρηπαίνουν περισσότερο την ατμόσφαιρα. Τι περιμένετε για να μην υπάρχουν άλλα diesel gates για να υπάρχει μια πραγματική έγκριση τύπου. Πρέπει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ανεξάρτητη ευρωπαϊκή αρχή που να κάνει την έγκριση αυτή και να ανακληθούν αυτομάτως ε, όλα τα οχήματα για τα οποία θα υπάρξει κάποια αμφισβήτηση για το κατά πόσο τηρούν ε, τους νόμους ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σούλτσε, δύο λεπτά. Κύριε Επιτροπέ, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή άρχισε τη λειτουργία της το Μάρτιο του 2016. Είχαμε ακροάσεις τεχνικών εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπροσώπων της αυτοκινητοβιομηχανίας, εκπροσώ... Ε, ακούσαμε επίσης και ε, ε, επιτρόπους και νομίζω ότι όλα πήγαν εξαιρετικά. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, θα πρέπει να αποφασίσουμε τι διατάξεις θέλουμε για τα επιβατικά οχήματα. Είναι σαφώς παράνομες, ε, όπως είπατε και εσείς, οι παράνομες αυτές διατάξεις, αυτοί οι μηχανισμοί αναστολής. Θα ε, πρέπει επίσης ε, να έχουμε και ακόμη να συνεχίσουμε να έχουμε αμφιβολίες για το αν μόνο η Volkswagen ήταν ένα δίκο. Αν δούμε και τις φήμες που που ε, κυκλοφορούν για τη Fiat, παραδείγματο χάρη είναι για άλλε εταιρείε, θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά ε, τι ε, ειδήσει που κυκλοφορούν. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι δοκιμέ οι οποίε γίνονται σε εργαστήριο. Θα πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα μέτρα τα οποία έχει ξεκινήσει η Επιτροπή. Μιλήσαμε και με τον Επίτροπο Ταγιάννη και με του άλλου επιτρόπου για τι νέε διατάξει. Η Επιτροπή έχει ακούσει πολλούς εμπειρογνώμονες και μηχανικούς και ε, θα πρέπει να φροντίσουμε οπωσδήποτε οι παράνομοι αυτοί μηχανισμοί αναστολής να ε, μην επιτρέπονται ώστε να επιτρέπεται η σωστή τεχνολογία ε, των δοκιμών. πολύ συχνά υπάρχει ε, η εντύπωση ότι ε, η Επιτροπή θέλει να αποδείξει ότι υπάρχει συνωμοσία μεταξύ Επιτροπής και αυτοκινητοβιομηχανίας. Ελπίζω όλοι να έχουν καταλάβει ότι δεν ισχύει αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Παολούτσι, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ, Μάσιμο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι εργασίε τη Επιτροπή Έρευνα έφεραν στο φω ξεκάθαρα πω το σκάνδαλο Volkswagen είναι μόνο η κορυφή ενό υπαγόγονου. Δεν είναι μόνο η απατελή χρήση δικών μηχανισμών για να λειτουργούν τα... οι κινητήρε με διαφορετικό τρόπο υπό διαφορετικέ συνθήκε. Ήδη από το 2011 ήταν γνωστό ότι τα αυτοκίνητα που τοποθετούνται στην αγορά και στην... Ε, στους κυκλοφορούν στου δρόμου έχουν εκπομπέ 7 με ε, φορές ψηλότερες από αυτές που δείχνουν οι εργαστηριακές δοκιμές. Μια τεράστια απάτη εις βάρος των πόλεων μας, εις βάρος ε, των ε, τρόπων, ενώ μάλλον υπάρχουν τεχνολογίες για να μειωθούν οι εκπομπέ των οξυδίων του αζότου. Γι' αυτό και θα πρέπει να αλλάξουμε τελείως του κανόνες για την πιστοποίηση, να ξεπεράσουμε και να επιβάλλουμε πιο αυστηρούς νόμους υπέρ της προστασίας των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζλωτόφσκι, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το σκάνδαλο ε, το οποίο οδήγησε στη δημιουργία αυτής της Επιτροπής Ερεύνης έχει επιβαρύνει, έχει μάλλον ε, μειώσει την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στις σμούς της Ένωσης. Βεβαίως τα δικαιώματα των καταναλωτών είναι αυτά που παραβιάστηκαν. Ωστόσο, Πρόκειται επίσης και για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ευρωπαϊκή αγορά ε, στις νέες ε, χώρες αλλά και στις χώρες μας. Δυστυχώς παρά τις πολυάριθμες ακροάσεις εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να κλείσουμε την έρευνα και να ορίσουμε αν επρόκειτο από πλευράς της Volkswagen για η θελημένη ε, απάτη. Ελπίζω πως αυτή η τελευταία φάση της Επιτροπής ε, ε, Ερεύνης θα δώσει τις απαντήσεις για το ποιος είναι αλλά θα πρέπει να αποφευχθεί η μόνιμη ύφεση για την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λόπες Βερμέχο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται σαν να είμαστε υπερβολικά προνοητικοί για άλλη μια φορά να μιλάμε για ένα πολιτικό συμπέρασμα όσον αφορά το κινητήρα diesel. Μα γνωρίζουμε ότι η ύπαρξη τέτοιων μηχανισμών αναστολής και η διαφορά όσον αφορά την ε, ρήπανση από τους νέους κινητήρες είναι πράγματα τα οποία ήταν γνωστά και κανένας δεν έκανε τίποτα. Στις αοκράσεις η Αυτοκινητοβιομηχανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, περνάνε από αντίφαση σε αντίφαση και δεν μπορούν να αρνηθούν ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες επηρέασαν τις αποφάσεις μας όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και δεν εφάρμοσαν τις ήδη υπάρχουσες υπέρ των δικών τους συμφερόντων. Η περίπτωση αυτή μπορεί να είναι όντως η κορυφή του παγόβουνου σε σχέση με το πώς καθορίζουν οι πολυεθνικές τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Παρόλο που είναι πράγματα τα οποία πειράζουν την καθημερινότητα των πολιτών μας. Έχουμε χιλιάδες πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο εξαιτίας των οξυδίων του αζότου. Αν μη τι άλλο, αυτά πρέπει να τα λέμε στην εκθεσή μας. 1,5 λεπτό, κυρία Ρέντα. Τζούλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε δει αρκετέ ε, λήψει όσον αφορά την ε, δημιουργία τη Επιτροπή, τη Εξεταστική Επιτροπή. Ε, αντίδραση τη Επιτροπή για την παροχή εγγράφων ήταν μία ικανοποιητική. Χρειάστηκε αρκετή καθυστέρηση στη συνεργασία μα και με το Κοινό Κέντρο Ερευνών υπήρχαν πολλές δικαιολογίες όσον αφορά το, τον όγκο των εγγράφων και πολλές φορές τα έγγραφα δεν ήταν τα κατάλληλα. Η Επίτροπος Μιανκόφσκα χθε εξέφρασε τη δική της δυσαρέσκεια με το κατά πόσο ε, τα κράτη-μέλη ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Κυρία Μιανκόφσκα, νομίζω ότι τώρα είναι η δική σα αρμοδιότητα να μας παρέχετε πληροφόρηση ε, με τρόπο πλήρη και άμεσο πρώην Επίτροπη αρνήθηκαν να εμφανιστούν στην Επιτροπή. Αυτό φαίνεται ότι ε, είναι αντίθετα με το άρθρο 198 που είναι το δικαίωμα των καταναλωτών να γνωρίζουν. Ευχαριστώ. Κύριε Στέφανε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η Εξεταστική Επιτροπή, εμείς, φτιάχτηκε για δύο λόγους. Πρώτον, για να καταλάβει για ποιο λόγο φτάσαμε στο σημείο όπου αυτοκινητοβιομηχανίες να παρακάμπτουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, πώς έγινε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος που φτιάχτηκε αυτή η Εξεταστική Επιτροπή ήταν να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων καταναλωτών στα προϊόντα μας. Το έργο της θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα στο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περισσότερο σαφή και να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με την πραγματικότητα. Πρέπει να αναγνωρίσω ότι πιστεύω πω κάποια πρόοδο έχει επιτευχθεί από τι συζητήσει μα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν μη τι άλλο, είπαμε ότι οι μετρήσει δεν πρέπει να γίνονται θεωρητικά, αλλά πρέπει να γίνονται στην πράξη πάνω στου δρόμου και να υπάρχουν ε, ίδιε προποθέσει για όλου. Όμω πρέπει να πω ανοιχτά ότι δεν συνεργάζονται όλες οι χώρες μέλη, πράγμα το οποίο καθυστερεί τη διαδικασία και την κάνει πιο περίπλοκη. Το θέμα αυτό βέβαια έχει και μία άλλη πλευρά, το ότι χιλιάδες ε, καταναλωτές εξαπατήθηκαν. Οι επιχειρήσει στην Αμερική πληρώνουν χιλιάδε δολάρια στους καταναλωτές, ενώ στην Ευρώπη αρνούνται να πληρώσουν οποιαδήποτε αποζημίωση. Αν θέλουμε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πρέπει να κάνουμε τα πάντα, ό,τι περνάει από το χέρι μα, ώστε και οι Ευρωπαίοι να αποζημιωθούν κατάλληλα και δίκαια για τη ζημιά που υπέστησαν και για τα ψέματα που του σερβίρανε. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, όχι να τιμωρήσουμε την βιομηχανία αλλά ε, γιατί και εκείνη προσπαθεί να εισάγει καινοτομία κτλ. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μη τι άλλο, πρέπει να δημιουργήσει ένα δίκαιο χώρο, ένα δίκαιο περιβάλλον για όλες τις επιχειρήσεις και να φροντίσει όλες να συμμορφώνονται προς τους κανόνες. Ευχαριστούμε κύριο Σερτούγκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Τι τελευταίες εβδομάδες ε, είδαμε ε, τις απαιτήσει που υπάρχουν από την Εξεταστική Επιτροπή. Από τις ακροάσεις μέχρι τώρα ε, μπορούμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στις ερωτήσεις μας ε, ακριβώς ε, με όσα χρειάζεται, αλλά όχι να μας πει, αλλά όχι με πλειέστατες ε, απαντήσεις. Η Επιτροπή φαίνεται να μην θέλει να έχει επίγνωση των εξουσιών τις οποίες διαθέτει. Επίσης, δεν είναι σαφές το πώς τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ή δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. η Επιτροπή ε, ε, ακόμη και για διατάξεις ψήξης ε, αυτοκινήτων είχε ένα μεγάλο κατάλογο με παραβάσεις τις οποίες μπορούσε να προωθήσει. Πιστεύω ότι και τα κράτη-μέλη έχουν μέρος της ευθύνης, αλλά μεγάλο μέρος της ευθύνης έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Ευχαριστώ. Κυρία Γκέρλινγκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους εισηγητές για αυτή την ενδιάμεση έκθεση. Δεν μας λέει και πολλά πράγματα, αλλά τουλάχιστον ε, παρουσιάζει την πορεία την οποία ακολουθούμε. Εγώ ήμουν ε, εισηγήτρια για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και γι' αυτό ήρθα σε αυτήν την εξεταστική επιτροπή. Στην αρχή της διαδικασίας, ε, πριν από τρία χρόνια περίπου, ξεκίνησαν τα προβλήματα και από μια παρουσίαση της Γενικής Διεύθυνσης ΕΝΒΗ είδα ότι κατάλαβαν πάρα πολύ καλά ότι δεν ε, ε, ανταποκρίνονταν οι προδιαγραφές με αυτά τα οποία ε, απέδιδαν τα οχήματα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Και ήμουν απόλυτα αποφασισμένη ότι πρέπει να φτάσουμε στην πραγματική αιτία των πραγμάτων. Σε αυτή τη συγκεκριμένη εξεταστική επιτροπή υπάρχουν και πολιτικά και τεχνικά θέματα. Αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει είναι να διασφαλίσουμε ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα ξέρουμε ποια είναι τα πολιτικά διδάγματα που πρέπει να πάρουμε, θα καταλαβαίνουμε πλέον πολύ καλά ποιοι φορείς, ποια, ποιες υπηρεσίες της Επιτροπής πρέπει να συνεργάζονται με τρόπο σωστό και άμεσο ε, και να λαμβάνουν τις ευθύνες του σοβαρά υπόψη και πώς θα εφαρμόσουμε ένα σύστημα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Νίτερ δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μάθαμε πολλά κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, όχι μόνο για τη Volkswagen, αλλά κυρίως για το πώς πρέπει να υλοποιείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία, πώς πρέπει να υπάρχει επιμερισμός ευθυνών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών και σχετικά με την δεοντολογία και την πρακτική ορισμένων εταιριών. Μάθαμε πολλά, τα οποία ήταν και πολύ απογοητευτικά. Έχουμε όμως την ευκαιρία να αλλάξουμε πράγματα για να τα κάνουμε καλύτερα. Η βιομηχανία πρέπει να έχει ξεκάθαρους κανόνες στους οποίους θα πρέπει να υπακούει και δεν πιστεύω ότι είναι πολύ ακριβά αυτά τα μέτρα και δεν μπορεί να τα εφαρμόσει η αυτοκινητοβιομηχανία. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο μέλλον γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό για τις εργασίες της Επιτροπής και θα πρέπει να κατανοήσουμε τα βασικά στοιχεία από τα οποία θα ήθελα να αναφέρω κάποια. Πιστεύω ότι μόνο τα οχήματα που σέβονται τους κανόνες θα πρέπει να επιτρέπεται ε, να διατίθεται στην αγορά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε διότι οι κανόνες θα πρέπει να τίθενται σωστά και ε, θα πρέπει να αποφεύγουμε περί τους κινδύνους για την ε, υγεία. Ε, ξέρουμε ότι με την υφιστάμενη τεχνολογία μπορούμε να έχουμε καθαρά οχήματα και στο μέλλον. Ε, δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα. Καθυστερήσαμε ε, στην εισαγωγή των καλύτερων εργαστηριακών δοκιμών. Τώρα θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να απαγορεύονται οι αλλοιώσεις μηχανισμών στα οχήματα κατά τη διάρκεια των δοκιμών στο μέλλον πρέπει να έχουμε καλύτερα συστήματα, να δίνουμε υποστήριξη ε, για τις δοκιμές και για ανεξάρτητες δοκιμές. Πιστεύω ότι τα σφάλματα μέχρι τώρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να έχουμε στο μέλλον ένα σύστημα καλύτερο για όλους μας. Και είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Σαλντεμόζε, ένα λεπτό. Κριστέλ. Πρόεδρε, το σκάνδαλο των μηχανισμών αυτών δεν είναι μόνο σκάνδαλο επειδή είναι απάτη, πρόκειται και για τον κίνδυνο των ανθρώπων που εκτίθενται σε αυτά τα οξύδια του αζότου που μάλιστα ε, ε, εκπέμφθηκαν ε, εξετέθησαν σε αυτά τα αερία οξύδια του αζότου ε, για τόσο χρόνο. 72.000 κόσμος πεθαίνει λόγω της ρήπανσης και οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και το περιβάλλον υποφέρει και στην Επιτροπή μας αυτό εξετάζουμε γιατί φτάσαμε σε μια τέτοια κατάσταση και γιατί δεν αποκαλύφθηκε αυτό το σκάνδαλο πολύ νωρίτερα. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα στο σύστημα. Ε, κανείς δεν θέλει βεβαίως να αναλάβει τις ευθύνες και ο ένας πετάει τον παλάκι στον άλλον αλλά εδώ θέλουμε να ελέγξουμε αυτά τα αυτοκίνητα που, που είναι προβληματικά. Το σύστημα ελέγχου μας θα πρέπει να είναι πολύ πιο ξεκάθαρο, να μην υπάρχει καμία πια αμφιβολία και να ξέρουμε επίσης και σαφώς ποια είναι η κοινή ευθύνη. Ας δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα για να προστατεύσουμε τον άνθρωπο και τη φύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Το και ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Οι συνεχιζόμενες εργασίες της Επιτροπής Ερεύνης δίνουν, δίνουν μια καλή εικόνα για τα τεχνικά συστήματα των κινητήρων ε, καύσης. Είναι ε, έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλές πληροφορίες για τεχνικές ε, πτυχές αλλά και για τις νομοθετικές διαδικασίες. Εγώ ε, προσωπικά πήρα το εξής δίδυγμα. Σχηρή πολιτική πίεση για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα οδήγησε σε απαράδεκτες διαδικασίες και σφάλματα τους κατασκευαστές όπως την Volkswagen και αυτό δημιουργεί πολύ, πολύ με τεράστιες δυσκολίες. Ε, τα αποτελέσματα της εργασίας της Επιτροπής θα μας δείξει τι και πώς λειτουργήσαν οι κατασκευαστές στη διάρκεια αυτής της θητείας, αλλά και πώς θα συντάξουμε καλύτερη και σωστότερη νομοθεσία που θα ορίζει τεχνικώς εφικτές εμ, όρους για τον έλεγχο αλλά και για την πιστοποίηση για τις άλλες χώρε. Ευχαριστώ. Γκαμπιού, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, τον Ιούλιο που μας πέρασε ομόφωνα εγκρίναμε την προσωρινή μας έκθεση. Τηρήσαμε δηλαδή την εντολή η οποία μας δόθηκε για το σκάνδαλο αυτό που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έπληξε χιλιάδες ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν την εξεταστική αυτή επιτροπή με εντολή συγκεκριμένη και σήμερα θέλουμε να εγκριθεί από την Ολομέλεια η έκθεση αυτή προκειμένου να συνεχίσει να προχωράει στο βάθος της υπόθεσης η Εξεταστική μας Επιτροπή. Σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα, πιστέψτε με. Οι ευρωβουλευτές εδώ που συμμετέχουμε και στις Επιτροπές Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε να συγκεράσουμε πολύ διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ τους. Η βιομηχανοποίηση της Ευρώπης απαιτεί μια στρατηγική που να προστατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, αλλά συγχρόνως να στοιχηματίζουμε και υπέρ της καινοτομίας και της βιομηχανίας και της καινοτομίας. Θέλουμε να ρίξουμε φως σε μια υπόθεση όπου δεν τηρήθηκαν οι κανόνες υπό τον Επίτροπο Φερχόγεν και από εκεί οδηγηθήκαμε στη σημερινή κατάσταση. Είναι δύσκολο βέβαια το έργο της Επιτροπής μας. Μην ξεχνάμε ότι ε, κάποιοι αρνήθηκαν να εμφανιστούν μπροστά στην Επιτροπή μας για ακρόαση. Σίγουρα όμως πρέπει να στραφούμε προς το μέλλον. Με, να ρίξουμε φως στην υπόθεση, με ταχυγράφους. Εμείς στρεφόμαστε λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΗΠΑ και όλες τις αρμόδιες αρχές και ζητούμε να συνεργαστούν και να τηρήσουν ε, την αρχή της ε, θεμητής συνεργασίας προκειμένου να βελτιωθεί το μέχρι τώρα έργο μας και να αποφύγουμε ε, νέα παραβίαση κανόνων. Διότι η προτεραιότητά μας είναι η υγεία των πολιτών, η ευημερία τους. Και έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε στο τέλος της αποστολής μας, να αποδώσουμε ευθύνε και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ενός ε, τομέα ο οποίος μέχρι το 2025 πρέπει να έχει δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστούμε πολύ, η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι, παιδιά, αρρωσταίνουν, χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας των υψηλών επιπέδων ρήπανσης της πόλης μας. Δεν βλέπουμε τίποτα καινούριο εδώ. Κανονικά πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες που να το απαγορεύουν. Όμως μέχρι σήμερα κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. Και δεν περιοριζόμαστε σε μια αυτοκινητοβιομηχανία πάνω από μια παράγει ε, ρήπους 10 φορές παραπάνω από ό,τι προβλέπουν οι προδιογραφές. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε συνενοχή των δημοσίων αρχών πια που καλύπτουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες που παραβιάζουν τους κανόνες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε μια τέτοια κατάσταση όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες να αισθάνονται τόσο άνετα όντας σίγουρες πως οι αρχές θα τους καλύψουν. Δεν πρέπει κανένας να νιώθει άνετα στην παρανομία. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τις, την εξεταστική μας επιτροπή, να καταλήξουμε σε συστάσεις ώστε τέτοια πράγματα να μην ξανασεβούν ποτέ. Ευχαριστούμε κύριε Ανταλή. Ο κύριος Φαντάλεν τώρα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλου όσοι βοηθάνε στην εξεταστική αυτή επιτροπή, η οποία έχει πάρει το δρόμο τη και όντω σιγά σιγά έχουμε περισσότερε πληροφορίε από όλου του εμπλεκόμενου. Όμω, κάποια στιγμή πρέπει να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και μετά τα συμπεράσματα να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα. Έτσι δεν είναι. Με ποιο τρόπο όμως θα πείσουμε τις κυβερνήσεις και την αυτοκινητοβιομηχανία όταν υπάρχουν χιλιάδες λόμπιστ, ομάδες πίεσης, οι οποίες επίτηδες ρίχνουν ε, καπνό στα πράγματα, δεν αφήνουν να δούμε καθαρά το τι συμβαίνει. Πώς θα καταφέρουμε να έχουμε αυτοκίνητα χωρίς ε, ρήπους. Υπάρχουν όμως καθαρά αυτοκίνητα, υπάρχουν καθαρά καύσιμα και χωρίς τέτοιους μηχανισμούς αναστολής. Προς τα πού πάμε. Η Ευρωπαϊκή Άνωση εκεί πρέπει να βάλει την ενέργειά της. Σε αυτά για να έχουμε αυτοκίνητα χωρίς εκπομπές. Κράτσια. Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή για την εργασία του. Με αυτή την έκθεση είναι μια καλή σύνοψη ενός εξάμεινου εργασίας στην Επιτροπή ΕΜΙΣ. Ωστόσο η εντολή μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες αλλά και πολλές, πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Όλοι εδώ προσβλέπουμε στα τελικά πορίσματα. Δεν μπορεί αυτό να γίνει χωρίς μια στενή και πιστή συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη διάρκεια των συνεδριάσεων πολύ κατηγορήσαμε την Επιτροπή επειδή δεν μπόρεσε να αναθεωρήσει τη διαδικασία έγκρισης τύπου και του ελέγχου. Όμως δεν είναι πλήρης αυτή η εικόνα. Όχι μόνο καθυστέρησε στην ανάληψη δράσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο έχασε χρόνο μέχρι ότου ολοκληρώσει την πρώτη του έκθεση όσον αφορά την, τον, την νομοθεσία περί ε, ελέγχου ε, εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες. Το τελικό ε, αποτέλεσμα ήταν ότι οι πελάτες έχασαν την εμπιστοσύνη τους στον ε, κατασκευαστή ε, των αυτοκινήτων και οι καταναλωτέ υπέφεραν από αυξημένη ατμοσφαιρική ρήπανση. Εμεί ε, ελπίζουμε ότι η Volkswagen θα αναγκαστεί από την Επιτροπή να αποζημιώσει όλου του πελάτε τη από τι παράνομε αυτέ τι πρακτικέ εντός τη Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τιμωρούν αυστηρά κάθε τέτοιου είδους πρακτικές. Κύριε Πρόεδρε, τώρα θα πρέπει να εστιάσουμε στο νομοθετικό έργο και να ολοκληρώσουμε την τρίτη και το τρίτο και τέταρτο πακέτο περί ελέγχου εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Θέλουμε να ολοκληρωθεί η τελική μας έκθεση, πράγμα που θα βελτιώσει το πλαίσιο εκπομπών από τα αυτοκίνητα. Ε, τώρα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η κακοδιαχείριση δεν θα ξανά υπάρξει. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε εδώ ώστε να προστατεύουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και καταναλωτές από τις απάτες. Ευχαριστώ κύριο Ζωγίνιο. Ένα λεπτό έχετε. Κάρλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων, της, της βιομηχανίας του, των πολιτών της Ευρώπης να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση προς την ευφυή κινητικότητα που βελτιώνει την ποιότητα ζωής και ανοίγει νέες προπτικές για ταγωνιστικότητα. Σε αυτό το τομέα η Επιτροπή ΕΜΕΣ είχε πολύ θετικό αντίκτυπο. Στη συνέχεια, μετά από αυτήν τα κράτη-μέλη και τα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να βγουν από τη ζώνη της άνεσής τους, να δουν πώς θα ελέγχουν καλύτερα, πώς θα διαδίδουν καλύτερα τη διαφανές και ξεκάθαρες πληροφορίες στους καταναλωτές και πώς θα φτιαχτεί το κοινό κέντρο ερεύνης. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι τεχνολογίες ελέγχου των εκπομπών εντός και εκτός Ένωσης ώστε να μην είναι πια ποτέ οι ίδιες. Εντόπιον ενδείξεων ε, ε, απατών, οι αρχές θα πρέπει να προβούν σε ένα τεχνολογικό άλμα. Είναι σημαντικό αυτό κύριε Επίτροπε, αλλά δεν αρκεί. Είναι σημαντικό να εκριζωθεί η νοοτροπία που επέτρεψε να συμβεί αυτή η απάτη. Αυτό το δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να ε, αναζητούμε διαρκώς. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Κυρία Γραπίνη, παρακαλώ Μάρια, θυμίζω ότι έχετε ένα λεπτό έκαστος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε, εξ αρχής ε, εκτιμώ αυτό το έργο αυτής της Επιτροπής στα μέσα της εντολής, αλλά θέλω να ε, υπογραμμίσω κάποιες, κάποια σημεία. Ακούσαμε στη διάρκεια αυτής της συζήτησης πολλά και διάφορα επιχειρήματα και συγκρίσεις ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την αποδοχή ανά, ανά τύπο ε, και διερωτώμε αν θα πρέπει να επιταχυνθεί η σύνταξη αυτής της έκθεσης ενώ αναμένουμε τα αποτελέσματα από την Επιτροπή. Όχι, δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε τα απορίσματα της Επιτροπής πριν να εγκριθεί αυτή η έκθεση και δεν νομίζω ούτε ότι στη ΣΥΠΑ λειτουργούν καλύτερα τα πράγματα από ότι εδώ ε, και έχουν πολύ πιο light ε, νομοθεσία και υπάρχει μια θελοντική συμμόρφωση. Προς αυτήν δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχουν απλοί νόμοι που προστατεύουν τον πληθυσμό χωρίς να δολοφονούν, να στραγγαλίζουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εγώ ε, προέρχομαι από τη βιομηχανία και έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές υπερνομοθετούμε και επιβαρύνουμε τις, επιτρο... τις ε, επιχειρήσεις, πράγμα που έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο. Και δεν είναι μόνο η Volkswagen, είναι και άλλοι κατασκευαστές που κάνουν λάθη σε αυτό το τομέα και πρέπει να μιλήσουμε για καθέναν από αυτούς. Ευχαριστώ. Σούλινγκ, ένα λεπτό. Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή εμείς, η Εξεταστική Επιτροπή, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τα θέματα αυτά. Συχνά λέγεται ότι υπάρχει πολύ κακή εποπτεία της αγοράς στην αυτοκινητοβιομηχανία και το σκάνδαλο της Volkswagen ήταν μια απόδειξη γι' αυτό. Οι μηχανισμοί αναστολή απαγορεύονται εδώ και χρόνια και παρόλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν. Φαίνεται ότι συνεχίζουν να υπάρχουν στους δρόμους ε, αυτοκίνητα με μηχανισμούς οι οποίοι είναι απαγορευμένοι. Θα πρέπει να αντιδρούμε με μεγάλη αυστηρότητα σε τέτοιου είδους σκάνδαλα και να επιβάλλουμε τις απαραίτητες κυρώσεις στους υπευθύνους παρά την απαγόρευση των μηχανισμών αναστολής φαίνεται ότι επιτρέπεται ακόμη να κυκλοφορούν τέτοια οχήματα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το συντομότερο δυνατόν. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να συνεργαστούν, διαφορετικά χάνουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η περίφημη ανταγωνιστικότητα των γερμανικών εταιριών οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις μίζες και στις παράνομες και βρώμικες πρακτικές που χρησιμοποιούν για να εξαπατήσουν τις ελεκτικές αρχές και τους καταναλωτές. Σε ερώτηση που κατέθεσα στις 23 Σεπτεμβρίου του 2015 είχα ζητήσει έρευνα που διεξήχθη στη ΣΥΠΑ και αποκάλυψε το σκάνδαλο της Volkswagen να επεκταθεί και στην Ευρώπη και να καλύψει και άλλες εταιρείες του κλάδου όπως επισημαίνει και η επίτροπος κυρία μπιενκόφσκα στην απάντησή της έρευνες που διεξήχθηκαν σε διάφορα άλλα κράτη μέλη απέδειξαν ότι υπήρξαν παραπτώματα και μέθοδοι καταστρατήγησης των αποτελεσμάτων και σε άλλους κατασκευαστές. θα πρέπει συνεπώς η ευρωπαϊκή ένωση να λάβει άμεσα μέτρα για την αυστηροποίηση των ελέγχων στα αυτοκίνητα όλων των εταιριών σε όλη την ευρώπη και να επιβάλλει βαρύτατες κυρώσεις σε όσους παρανομούν εύχομαι η νεοσύστατη επιτροπή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου να ρίξει άπλετο φω στι παράνομε πρακτικέ τη αυτοκινητοβιομηχανία το γρηγορότερο και να σεβαστεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. στι 2 μαρτίου του 2017 οι πολίτε πρέπει να γνωρίζουν. ευχαριστώ. Σε αυτή τη φάση πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μια συλλογική αποτυχία. Αποτυχία από πλευρά όσων προσπάθησαν να εξαπατήσουν με ειδικέ συσκευέ του πολίτε, την Κομισιόν και τα κρατημέλη γιατί αποκαλύφθηκε η απάτη. Αποτυχία της Κομισιόν, γιατί γνωρίζοντας, όπως είπε κάποιος επίτροπος, ότι οι κανόνες ήταν ελαστικοί και έτσι τους ερμήνευε και ο, η αυτοκινητοβιομηχανία, δεν ε, πρότειναν νέους κανόνες, νέες ρυθμίσεις, ώστε να αποφύγουν τη, τέτοιου είδους ε, γεγονότα. Και από την άλλη πλευρά και αποτυχία των κρατών μελών, γιατί οι εθνικές αρχές έχουν ε, το καθήκον να ελέγχουν και να διερευνούν ε, τις καταστάσεις ώστε τέτοιου είδους ε, περιστατικά τα οποία βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών να μην συμβαίνουν. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε ώστε στο μέλλον τέτοιου είδους πράγματα να μην επαναληφθούν. Μιλάμε για την υγεία μας, μιλάμε για το περιβάλλον αλλά και για την ε, αυτοκινητοβιομηχανία που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και τέτοιου είδους ε, απάτες δεν ωφελούν καθόλου ούτε την αυτοκινητοβιομηχανία που ε, απέναντι στην οποία δημιουργείται καχυποψία. Ευχαριστώ, Χωσέ Μάισνερ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή ε, έχει κάνει ε, ε, πολλά τα οποία θεωρώ θετικά και ίσως έχει και κάποια ελλείμματα. Η Volkswagen καταφέρνει να επιτύχει τα 80 μιλιγκράμμ στην Καλιφόρνια διότι εκεί υπάρχουν κυρώσεις και οφείλει να το επιτυγχάνει. Στην Ευρώπη φαίνεται ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για τη Volkswagen και υπάρχει μεγαλύτερος παράγων ανοχής. Αντί για 80 μιλιγκράμμ είναι τριπλάσια ε, η επιτρεπόμενη ε, εκπομπή. Θα πρέπει λοιπόν να εξαγάγουμε τα διδάγματα από αυτό ε, το γεγονός. Είναι σημαντικό λοιπόν όχι μόνο για τα αέρια του θερμοκηπίου και για το διοξείδιο του άνθρακος αλλά και για το οξύδιο του αζότου να έχουμε νομοθεσία η οποία θα είναι ρεαλιστική, θα επιβάλλει στην αυτοκινητοβιομηχανία αυτά τα οποία πρέπει να κάνει και βεβαίως θα πρέπει να ελέγχουμε με σωστή εποπτεία και το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να έχουμε και τα σύστημα ελέγχου εκπομπών πραγματικής οδήγησης. Ευχαριστώ πολύ. Νικόλα Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές φορές ε, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγηθεί στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Αρκεί κανείς να σκεφτεί τα αποτελέσματα της, ε, του Παρισιού και του αγώνα που κάνουμε τώρα στον ΙΚΑΟ ε, για την αεροπλοεία. Όμως εδώ αυτή η Επιτροπή που έχει φτιάξει το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα γιατί ο κόσμος έτσι δεν θα μπορεί να πει ότι η Ευρώπη πρώτη και καλύτερη παραβιάζει τους ίδιους τις νομοθεσίες. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να καταγγείλουμε αν αυτό φανεί απαραίτητο και τις ε, ε, τις ε, παραβατικές εφαρμογές της νομοθεσίας ακόμα και για αυτούς τους μηχανισμούς. Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται και σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτήν την έρευνα. Ευχαριστώ. Κούν ένα λεπτό κι εσείς. Κύριε Σκούν, ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν καταφέρουμε να έχουμε καθαρά οχήματα στους δρόμους μας, είτε με ε, ηλεκτρισμό είτε με υδρογόνο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα κατάσταση και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις ούτως ώστε και για τα οξύδια του αζότου και για το διοξίδιο του άνθρακος να τηρούνται οι νόμοι και οι διατάξεις ε, για τα όρια εκπομπών και θα πρέπει να υπάρχει σωστή εποπτεία ε, ούτως ώστε να ε, μπορούν να εγκατασταθούν οι διατάξεις με βάση ε, τις προδιαγραφές Euro 6 ούτως ώστε να μπορούν και οι αυτοκινητοβιομηχανίε να τηρούν τα 80 μιλιγκράμμα ένα χιλιόμετρο, ε, πράγμα το οποίο δεν κάνουν στην Ευρώπη, ενώ στην Αμερική καταφέρνουν να τηρούν τα 50 μιλιγραμμ ανά μίλι. Χρειαζόμαστε λοιπόν τις σωστές διατάξεις και τις, ε, τη σωστή τεχνολογία, ούτως ώστε οι ε, επιβλαβείς εκπομπές να μετατρέπονται σε ε, αέρια τα οποία δεν είναι επιβλαβή για την δημόσια υγεία. Αυτό θα πρέπει να μπορούμε να το ελέγχουμε με σωστές δοκιμές και με δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης έχοντας ε, ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει με 150 ή 170 ή 200 χιλιόμετρα την ώρα γιατί αυτό έχει τεράστια ε, διαφορά στο, στις εκπομπές. Περιμένουμε ε, το νέο σύστημα για εκπομπές σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης να το έχουμε μέχρι το 2017. Θα πρέπει αυτό να θέσουμε ως στόχο διαφορετικά στις πόλεις μας θα έχουμε συνθήκες οι οποίες θα είναι επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία και για το κλίμα. Επειδή όλοι οι συνάδελφοι ήταν ε, πολύ καλοί μαθητές, ε, κερδίσαμε χρόνο. Είμαστε μπροστά. Μήπως θέλει κανείς ακόμα να πάρει το λόγο? Όχι. Ωραία. Τότε λοιπόν θα πάρει το λόγο η Επίτροπος Μπιανκόφσκα. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τους αξιότιμους ευρωβουλευτές για τις παρεμβάσεις σας και για την ειλικρινή συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας. Σίγουρα ο στόχος είναι κοινό. Πρέπει να αποκαλύψουμε τα πάντα σχετικά με το σκάνδαλο των μηχανισμών αναστολής ελέγχων και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και να συνεχίσουμε και μετά με μέτρα. Φυσικά η διαδικασία πρέπει να διέπεται από διαφάνεια για όλους μας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι θα κάνω ό,τι χρειάζεται, ό,τι είναι αναγκαίο. Η εντολή της Επιτροπής καθορίζεται ως ε, θεματοφύλακα των συνθήκων προκειμένου να φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες και από την αυτοκινητοβιομηχανία. Αλλά εγώ δεν θέλω να παίξω το παιχνίδι που παίζουμε τώρα, δηλαδή να δαχτυλοδειχθώ τον έναν τον άλλον. Όχι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορώ 100% να τα βάλουμε όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες γιατί δεν έχουμε τη βεβαιότητα 100%. Υπάρχουν πολλές επιστολές που στέλνω συνέχεια προς τις χώρες ε, μέλη πιέζοντάς τους να μου δώσουν απαντήσεις. Αλλά δεν έχω όλες τις απαντήσεις και δεν έχω άλλου είδους νομική εξουσία στα χέρια μου. Πολλοί είπαν ότι πρέπει να προχωρήσουμε στις ανακλήσεις, αλλά ακόμα δεν γίνεται σε μερικές χώρες, έχουμε δει ότι προχωρούν ε, σε υποχρεωτικές ανακλήσεις, σε άλλες δεν εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι χώρες μέλη σιγά σιγά αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε καλύτερες πρακτικές, ότι πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια, ότι πρέπει να μας δίνουν όλες τις πληροφορίες τεχνικές και άλλες που χρειαζόμαστε η δέσμευσή του είναι εκείνη η οποία θα βοηθήσει να γίνεται καλά ο έλεγχος της αγοράς. Τώρα χρειάζομαι τη δέσμευση των χωρών μελών, όπως και τη δικιά σας βέβαια, ότι θα μπορέσουμε να εγκαθιδρύσουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο για τον έλεγχο των οχημάτων και θέλω να είμαι σαφής ότι αυτό δεν θέλω να το κάνω σε βάρος της αυτοκινητοβιομηχανίας καθόλου. Είμαι που είμαι υπεύθυνη για την βιομηχανία, οπότε θα κάνω ό,τι χρειάζεται προκειμένου να ανθίζει η αυτοκινητοβιομηχανία, να είναι ανταγωνιστική, αλλά προς το συμφέρον της βιομηχανίας σήμερα και πιστεύω ότι και η βιομηχανία αρχίζει να το καταλαβαίνει αυτό, πρέπει να είμαι αυστηρή, πρέπει να είμαστε αυστηροί και απαιτητικοί μαζί τους. Αυτή την κρίση θέλω να τη χρησιμοποιήσω και ελπίζω να είναι κοινό μα στόχο προκειμένου να έχουμε καλύτερη νομοθεσία, πιο αποτελεσματική, πιο αποτελεσματικού ελέγχου τη αγορά και δομέ. Και τη βιομηχανία να την κάνουμε να, κυκλοφο... να προχωρήσει προ την πορεία ε, πιο αποτελεσματικών ε, ελέγχων, πιο, καθαρών, ε, πιο καθαρού αέρα. Είναι πράγματα τα οποία είναι προ το συμφέρον όλων μας η στήριξή μας προς την αυτοκινητοβιομηχανία θα την βοηθήσει να πετύχει τους στόχους αυτούς. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Τώρα είναι η ώρα για να φροντίσουμε για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε και τώρα θα απαντήσουν οι δύο εισηγητές. Παύλο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ όλους για τόσα είπατε. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Κεμπράντη για τη συνεργασία που έχουμε μαζί και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί και στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης αυτής. Κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι δεν υπάρχει αρκετή φιλοδοξία και περιεχόμενο στην έκθεσή μου. Όμως υπενθυμίζω ότι πρόκειται για μια προσωρινή έκθεση και ότι αποφασίσαμε ότι θα είναι μια έκθεση καθαρά τεχνική. Ο κύριος Ντανξίγκη είπε ότι δεν πρέπει να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Συμφωνώ. Οι πολίτες δεν είναι αυτό που περιμένουν από εμά να τσακωνόμαστε χωρίς να πετυχαίνουμε καμία αλλαγή. Αντίθετα, πρέπει μαζί να καταφέρουμε να μάθουμε την αλήθεια. Και τι είναι πιο σημαντικό. Αυτό μαζί να κάνουμε προτάσεις προκειμένου να μην επαναληφθεί το ίδιο στο μέλλον. Έτσι λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή δεν μπορεί να είναι μια έκθεση σε βάρος της βιομηχανίας, δεν μπορεί να είναι μια έκθεση σε βάρος της απασχόλησης, καθ' άλλο. Πρέπει να είναι μια έκθεση υπέρ του περιβάλλοντος, μια έκθεση υπέρ της αυτοκινητοβιομηχανίας και μια έκθεση υπέρ της απασχόλησης. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ο κύριος Γκερμπράντη τώρα, ο συνεισηγητής και εσείς ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πως αυτή... Ε η συζήτηση δεν αφορούσε τόσο την διάμεση έκθεση, γιατί αυτή ήταν περιορισμένη στις διαδικασίες, σε διαδικαστικά θέματα. Περισσότερο αφορούσε την κατάσταση προόδου της ε, ε, Επιτροπής Ερεύνης μας. Γιατί πιστεύω ότι ήταν πολύ ενθαρρυντικά τα λόγια σας, διότι διαπίστωσα πολύ ε, κοινή κατανόηση για το πρόβλημα. Ότι δηλαδή δεν οδηγηθήκαμε σε κοινά συμπεράσματα απαραίτητος. Αυτή θα είναι και η πρόκληση για τον αγαπητό συνάδελφο Παύλο Στάλμπα και εμένα για το, να φτάσουμε σε κοινά συμπεράσματα τελικά. Αλλά πιστεύω πως είμαστε σε σωστό δρόμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε την... Ε, Έρευνα που συνεχίζεται. Έχουμε πολλά ακόμα να διερευνήσουμε και πολλά στοιχεία να βρούμε. Έχω, θέλω να τονίσω δύο στοιχεία. Πολύ ωραία τα είπε ε, Πολύ, με μεγάλη φράδια υπόθηκαν οι μυριάδες ευθυνών. Κανείς φαίνεται να μην είναι όμως τελικά υπεύθυνο στο τέλος. Ε, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε τα κρατημέλη, ούτε οι Εθνικές Αρχές, κανείς. Αυτό ίσως είναι ο πυρήνας του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και είμαι βέβαιος ότι όταν θα το ψάξουμε περισσότερο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα ε, που δεν θα δικατοπτρίζουν μόνο αυτήν την, αυτόν τον βιομηχανία αλλά και άλλου τομείς τη πολιτική επίση. Ο συνάδελφος Ιβο Μπέλετ είπε πως αν εξετάσουμε τι ευθύνε, πολλά έχουν να κάνουν με την ανικανότητα των κρατών μελών να αναλάβουν ευθύνε. και πιστεύω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί είπαν ότι πρέπει να καταδείξουμε ευθύνες, αν θα πρέπει ή όχι. Ε, πολιτική λογοδοσία είναι πολύ σημαντική και αυτό μπορεί να σημαίνει και το να ε, κατονομάσουμε τους υπευθύνου. Δεν είναι αυτό το οποίο προσβλέπω, αλλά είναι αυτό κομμάτι μιας ισχυρής δημοκρατίας και αυτό εξακολουθούμε να προσπαθούμε να φτιάξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνεχίσουμε σε αυτή την ε, πορεία. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, τους εισηγητές, την κυρία Επίτροπο ε, για αυτή την εις συζήτηση. Ε, η συζήτηση θα συνεχιστεί ε, συγγνώμη, η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα και θα ε, ξαναρχίσουμε τη συνεδρίασή μας στις 12.30.